Παρακαλώ, καθίστε όλοι. Πάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που είναι η συμφωνία σύνδεσης ή σύμπραξης για την Αγγλία. Παρακαλώ καθίστε και μην κάνετε θόρυβο. Θα σας παρουσιάσω επομένω το θέμα και κατόπιν θα δώσω το λόγο, επειδή είμαστε στο σημείο 4, ξαναλέει ο Πρόεδρος, που είναι η ψήφιση της Ελληνικής Συμφωνίας για τον ε, τομέα του κλάδου της Αλίας μεταξύ Ένωσης και Γουινέας. Αυτά τα οποία συζητήσαμε και συμφωνήσαμε χτες. Θα σας δώσω το λόγο όμως. Ήδη το θέμα συζητήθηκε χτες. Σας δίνω το λόγο απλώς για διαδικαστικό. Αν δεν πρόκειται για διαδικαστικό, όχι. Γιατί τα είπαμε, τα είπαμε εξαντλητικά. Άμα ξαναρχίσει η κουβέντα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, η παρέμβαση μου νομίζω ότι είναι όντως σχετική με το θέμα αυτό. Το προηγούμενο ήταν ένα θέμα ε, που θεωρητικά θα έπρεπε να μας επιτρέψει να θέσουμε ερωτήσεις. Δεν μπορέσαμε να θέσουμε ερωτήσεις και είναι πιστεύω σημαντικό να μπορέσουμε να παρέμβουμε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αυτό που έχω να πω σχετίζεται με την ψηφοφορία. Από τις πληροφορίες λοιπόν που λάβαμε σήμερα ακόμα δεν τροποποιούνται επαρκώς, δεν τροποποιείται επαρκώ το πλαίσιο ενώπιον του οποίου ε, έχουμε βρεθεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπερψηφίσουμε την, την ε, πρόταση σήμερα. Αφού λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ε, αλλάζει ουσιαστικά το πλαίσιο, και δεδομένη της σοβαρότητας της κατάστασης στη Γουινέα, αφενός και της αβεβαιότητας που επικρατεί, της ε, ασάφειας που επικρατεί για το μέλλον, προτείνω να μην ψηφίσουμε σήμερα. Σας διακόπτω γιατί είπα. Σας δίνω το λόγο για διαδικαστικό. Δεν διαδικαστώ αυτό που μας λέτε. Συγγνώμη, συμπαθάτε με. Εγώ προεδρεύω. Και σας το είπα ξεκάθαρα μόνο για διαδικαστική. Μα πρόεδρε, προτείνετε ψηφοφορία. Εγώ προτείνω διαδικαστικά να μην ψηφίσουμε σήμερα και εξηγώ τους λόγους μου. Υπάρχουν επαρκείς, θεμητοί, σοβαροί λόγοι έτσι ώστε να μην ψηφίσουμε σήμερα. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν είναι ο λόγος της διαφωνίας μας. Λόγος διαφωνίας μας είναι οι σημερινές συνθήκες, συνθήκες που επικράτουν. Αυτές με οθούν να προτείνω να μην ψηφίσουμε σήμερα. Και αν επιμείνετε, δεν θα συμμετάσχουμε στην ψηφοφορία. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να λάβει χώρα ψηφοφορία στην τωρινή κατάσταση. Όχι ότι δεν ε, ε, συμφώνουμε επί τη ουσία ή όχι και επιπλέον δεν βρίσκω καμία συνοχή προ αυτά που προτείνει η οχι και επιπλεον δεν βρισκω καμια συνοχη προς αυτα που προτεινει η επιτροπη Είμαι η Πρόεδρος, αναλαμβάνω την ευθύνη. Είπαμε, ψηφίζουμε σήμερα, εκτός εάν πρόκειται περί της πλειοψηφίας, αλλά βλέπω δύο-τρει το ζητάτε να μην γίνει. Επομένως, θα ψηφίσουμε και σας το λέω για να είμαστε ξεκάθαροι. Σήμερα είπαμε ότι θα ψηφίσουμε διότι δεν υπάρχει ο χρόνος ούτως ώστε να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας, τις δεσμεύσεις μας. Και εγώ φέρω αυτή την υποχρέωση για να μπορέσουμε να πάμε στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Υποχρεωτικά επομένω πρέπει σήμερα να γίνει η ψήφιση. Μιλάει ταυτόχρονα, κύριε Φεράρα, δεν σα έχω δώσει το λόγο. Εγώ δίνω το λόγο εδώ πέρα. Μιλάει ταυτόχρονα ο κύριο Φεράρα, δεν ακούγεται. Παρακαλώ, συμπεριφερθείτε όπω πρέπει. Είπαμε, εγώ διευθύνω τη συζήτηση. Το συμφωνήσαμε χθε. Έγιναν οι εξηγήσει όλε. Είχατε την ευκαιρία όλοι να λάβετε το λόγο και υπάρχει επίσης η έσχατη κρίση ας πούμε που θα είναι όταν κατέβει αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια. Να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Και αν μεταξύ σήμερα και της μέρα εκείνης της Ολομέλειας ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ξέρουμε ότι ε, μπορεί κανείς να υποβάλει ένσταση εν ώψη της Ολομέλειας. Όμως θα είμαστε προετοιμασμένοι. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Από αυτή την υπόθεση εξαρτώνται πολλά χρήματα, μεγάλες ενισχύσεις. Άρα, γι' αυτό σας λέω. Δεν θα τα στο λόγο και πάμε τώρα να ψηφίσουμε. Όποιος δεν θέλει ας κάτσει και να απόσχει. Πάμε να ψηφίσουμε. Όχι, δεν θα σα δώσω το λόγο γιατί ανοίγει εκ νέου συζήτηση. Και ψηφίζουμε. Είσαστε ελεύθεροι να ψηφίσετε υπέρ, κατά ή να απόσχετε. Ψηφίζουμε. Τροπολογία περιθμών 1. Η συγκήτρια. Τι θέλετε συγκήτρια, θέλω να είμαστε λέει. Έξι ζητούν ονομαστική. Έτσι, έτσι απαιτείται. Ιδάλλως δεν γίνεται. Πολύ ωραία. Ωραία, θα γίνει ονομαστική ψηφορία επομένω. Ε, Some members don't have their cards. say, well, no, this is not the problem. I mean, if they don't have the cars, they don't have the cars. ¿Eh? Sometemos a votación y propongo, porque creo que hay diputados. Ωραία, θα ψηφίσουμε. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτέ που δεν έχουν την κάρτα. Οπότε Εάν δεν έχετε αντίρρηση, να γίνει έτσι. Ψήφισμα τώρα τροπολογία υπαριθμών 1. Αφορά το άρθρο 3α. Ψηφίζουμε. Ναι, sistema. καλμα, calma, calma, calma, calma, <laughs>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 que lo que se ha pedido el voto nominal es en Τροπολογία, της Ποιοι είναι υπέρ. Δεν είναι κράτα σημειώσεις για Ποιοι είναι κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της Ποιοι είναι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 της Επιτροπής των Προπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 2 των Προπολογισμών. Τροπολογία υπαριθμών 1 της Επιτροπής των Προπολογισμών. Υπέρ. Ξαναλέει πρόεδρος. Μετρήστε, μετρήστε τις ψήφους υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 2 της Επιτροπής των Προπολογισμών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται υπαριθμών 1 και άρα καταπίπτει υπαριθμών 3. Στη συνέχεια. Πάμε στην υπαριθμόν 5 της Επιτροπής Ανάπτυξης. Υπέρ. Κατά. Παρακαλώ, μετρήστε, κάντε την καταμέτρηση. 5. Επιτροπή Ανάπτυξης. Υπέρ. 9 εννέα, δέκα, απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω, ψήφι, υπέρ, για το 5 Μετρήστε, μετρήστε. Να, γιατί βλέπετε εδώ πέρα Έχουμε για άλλους ύπου που δεν Να εδώ στο πρόεδρο. Καφέ σύμπλε. Ψήφι κατά, εάν τέλειωσε. Εάν τέλειωσε.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 να μετρήσω. Κάποιοι δεν ψήφισαν πριν, ψηφίζουν τώρα, δεν ε, γίνεται καταμέτρηση. Τι να σου πω, κάντε θέλετε. Όχι, όχι, όχι. Έγινε λάθος. Έγινε λάθο. Ε, στην καταμέτρηση, λέει ο κύριο Μιλάνα, να αλλάξουμε αυτόν που κάνει την καταμέτρηση. Ας αντικαταστήσει κάποιον ε, το, το, γραμματεία που μετρανεί. Ωραία. Εάν δεν δουλεύει το μηχάνημα, λέει ο πρόεδρο, τότε θα πρέπει κάποιο. Τι θέλετε. Έχετε το λόγο, κύριε Ρώτη. Α κάνουμε τελική ψηφοφορία και να κάνουμε εκεί πέρα την επαλήθευση. El único problema no votamos la resolución legislativa quiere decir que da igual lo que hemos Έτσι δεν προχωράει το θέμα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα αν δεν κάνουμε την ψηφοφορία. Ναι, ναι, θα ψηφίσουμε. Σα είπα ότι αν δεν ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα δεν θα γίνει η ψήφιση στην Ολομέλεια. Αυτό το είπαμε, δεσμευτήκαμε και θα γίνει. Και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση της ε, Επιτροπής όπως έχει τροποποιηθεί. Ψήφι υπέρ. Ονομαστική είπαμε, αλλά δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Άρα θα πρέπει ένας ένας να καλείται και να ψηφίσει γιατί δεν λειτουργεί το μηχάνημα, δεν μπορώ να το φτιάξω. Ωραία, ας θα γίνει τότε λοιπόν κλίση ονομαστική, αφού θέλετε. Στίβενσον, Κάντικ, Μιλάνα,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 A ver, por favor, les pido calma porque ya... Παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία γιατί ήδη αρκετά μπερδεμένα τα πράγματα. Κύριε Αντίνορα, και πάλι. Πετε μα, ναι. Sí. Señor Iturgaiz, señora Patrao, señor Rivellini, señor Valesa, señor Andrés Barea, señor Arsenis, no está, eh, se, señora Yotova,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 ξαναμετράμε, να δούμε αν έχουν ψηφίσει όλες οι πολιτικές ομάδες. El resultado del voto de la propuesta de... Το αποτέλεσμα της ψήφισης για την πρόταση της ε, ευρωπαικη επιτροπης Επιτροπής είναι ότι έχουμε 15-3 με μία εποχή. Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε εποχή, διορθώνει ο γραμματέα. Ε, ε, por tanto, por mayoría queda aprobada la propuesta. Επομένω, με αυτή την πλειοψηφία εγκρίνεται η τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα θα ψηφίσουμε νομοθετική πρόταση και πάλι αρχίζουμε ε, αν την ώρα. Αρχίζει η εκφώνηση από την Πρόεδρο, την ονομαστική ψηφοφορία. Sí. Señor Iturgaiz, señora Patrao, señor Rivellini, señor Valesa, eh, señor Andrés Barea, eh, señor, eh, señora Aitoba,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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, no, no, no, no. Complet. Vamos a volver a repetir entonces. Cadec. C'est moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. 6. Y no, hay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 Όλο αυτό για τίποτα. Αυτά. Και έτσι ολοκληρώθηκε μετά της ψηφοφορίας. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα τη σημερινής διάταξης. On va faire les listes après, parce que c'était par rappel. Pasamos al punto siguiente del orden πάμε στο επόμενο θέμα τη μέσης διάταξη. Πρόκειται για το υπαριθμό 12, δηλαδή το οποίο αφορά το Συμβούλιο Αλίας για την Μεσόγειο και τις σχετικές διατάξεις που θα πρέπει να μεταφερθούν στο κοινωτικό δίκαιο. Παρακαλώ, μπορείτε να πάτε έξω από τον διάδρομο. Έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. El ε, señor Shali. El ε, señor Shali, por favor, le pido que tome la palabra para presentar la propuesta. Παρακαλώ, μπορείτε να μα προσθέσετε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει Επιτροπή. Por favor, pido Παρακαλώ, δείξτε σεβασμό στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει να λάβει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ονομάζομαι Τζούλις Λάγκεντορφ. Είμαι ε, αναπληρωματικός τμήματάρχης, υποδιευθυντής του τμήματος για την ε, ΛΙΑ και θα σας παρουσιάσω το σημείο 11, την προετοιμασία για την ένταξη στο παράρτημα 1 του τους ΣΥΤΕΣ. Έχουν γίνει κάποια βήματα μέχρι στιγμής. Να σας κάνω μια σύντομη αναδρομή, ιστορική αναδρομή και μετά να σας περιγράψω τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Όπως ε, θα γνωρίζετε, έχει υπάρξει προσέγγιση για το, στο ΣΥΤΕΣ ε, από το Μονακό και έχει ρωτήσει κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν όλα αυτά να αντιστοιχίσουν στην ε, αίτηση του, να συμφωνήσουν μάλλον στο αίτημα του Μονακό για την ένταξη στο παράρτημα 1 της σύμβασης ε, ΣΥΤΕΣ. Ε, αυτό έγινε τον Ιούλιο και η Κομισιόν έκτοτε είχε κάνει μια εκτίμηση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται, εκτίμηση δηλαδή για τις διαφορετικές προτάσεις που υπάρχουν για την COP15 του ΣΑΙΤΣ που θα γίνει το Μάρτιο του 2010 και εδώ έχει προσθεθεί και η πρόταση του Μονακό για τον ερυθρό τόνο. Αυτό περιλαμβάνεται στο έγγραφο εργασίας της Κομισιόν, το οποίο θα πρέπει να έχετε δει. Δημοσιεύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου. Μετά από αυτό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, έγινε μια συζήτηση για τις διάφορες προτάσεις και το, πρόγραμμα εργασίας της, το, το έγγραφο εργασίας της Κομισιόν προς την Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΥΤΕΣ. Έγινε μια σχετική συνεδρίαση στις 21 Σεπτεμβρίου. Ε, την περασμένη εβδομάδα όπου η αξιολόγηση της Κομισιόν για την πρόταση του Μονακό συζητήθηκε και το τελευταίο, τελικό αποτέλεσμα αυτής της συνεδρίασης περιλαμβάνεται στην σύνοψη των συμπερασμάτων που ε, υπάρχει διαθέσιμη, είναι δημόσια διαθέσιμη και εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες. Τώρα, τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν σε σχέση με τη διαδικασία είναι ότι εάν το Μονακό επιμείνει στην πρότασή του, θα πρέπει να υποβάλει την πρόταση στο site στο παράδειγμα 1, μέχρι την 4η Οκτωβρίου. Αυτή είναι η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για την COP15 και μετά από αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα εφόσον η απόφαση λήφθη ότι είναι πρόημο η κοινότητα να υποστηρίξει την πρόταση του Μονακό σε αυτή τη φάση. Αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν προκαταλαμβάνει την θέση που τελικά θα κρατήσει η Επιτροπή στις περαιτέρω φάσεις, δηλαδή ανάμεσα στις 14 Οκτωβρίου αν το Μονακό καταθέσει αυτή την πρόταση επισήμως και την διεξαγωγή της COP15. Οι συζητήσεις που θα γίνουν θα γίνουν επί τη βάση μιας πρότασης της Κομισιόν για απόφαση από το Συμβούλιο επί τη βάση του άρθρου 322 της συνθήκης και θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της ετήσιας συνεδρίασης της ΆΙΚΑΤ που θα γίνει τον Νοέμβριο του 2009. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ποια είναι τα διαδικαστικά ε, βήματα και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ε, ε, πολύ ωραία. Δεν μα διαφωτίζεται και πάρα πολύ σχέση με τη διαδικασία, αλλά τέλο πάντων, Ρωμέρα, για το λόγο. Ακριβώ, ακριβώ θέλω το λόγο, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει κάπω περισσότερο να σταθούμε στη διαδικασία. Να σα πω τι σκέψει μου. Πρώτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσουμε το τι προηγήθηκε αυτή τη απόφαση του Μονακό. Γιατί όταν στο Μονακό προτείνεται να ε, πάει στο πρώτο παράρτημα ο κόκκινο τόνο είναι γιατί έχουμε όλου αυτού του μηχανισμού που έχουν προταθεί για να σώσουμε αυτό το ψάρι που απέτυχαν ή δεν εφαρμόστηκαν ή από πλευρά συλλεκτικών μηχανισμών υπάρχει πρόβλημα. Δεν λειτουργήσε το σύστημα και επομένω τελική συνέπεια ήταν ότι καταλήξαμε στο ΣΥΤΕΣ. Αλλιώ ε, έτσι δεν έγινε με κάποιο άλλο τρόπο αυθόρμητο και εκ των ενόντων γιατί στο προηγούμενο πριν από αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και έτσι έχουμε αχθεί σε αυτή τη λύση και τώρα θα πρέπει να εξελογήσουμε για να δούμε αν είναι τώρα ή όχι η κατάλληλη στιγμή ε, γιατί και στην ΙΚΑΝΤ είχε συζητηθεί αυτό, είχαν υπάρξει προτάσεις ε, επιστημονικές οι οποίες τελικά δεν υιοθετήθηκαν ή τουλάχιστον ε, όχι στο δέν μέτρο. Μην το ξεχνάμε αυτό, διότι τώρα γίνεται αυτή η συζήτηση και θα γίνει και στου μέσο επόμενο μήνε πριν από το ΙΚΑΤ και πριν την τόχα του του Μάρτη και θα είναι πάρα πολύ βασικό το τι θα πούμε. Αν τώρα αναβληθεί η απόφαση αυτό σημαίνει ότι, ότι η πρώτη μου ερώτηση είναι αυτή, εάν επομένως η Κομισιόν αναβάλει τότε Πάρα πολύ δύσκολο να ζητηθεί αυτό το πράγμα το Μάρτιο στην ε, Ντόχα. Δύσκολο να μπει στη μέση διάταξη. Άρα, είναι τώρα η στιγμή ή δεν είναι. Αν είναι και αν είναι αργότερα, εσείς με τι χρονοδιάγραμμα βλέπετε ότι θα μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Άλλωστε, η ΣΥΤΕΣ δεν συνεδριάζει κάθε μήνα. Άρα, για πέστε μας, εάν όχι τώρα, πότε είναι η επομένη ευκαιρία για να συζητηθεί το θέμα. Αυτό είναι το πρώτο μου θέμα. Το δεύτερο τώρα. Έχει υπάρξει μια εξέλιξη στα θέματα αυτά. Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, ε, Γερμανία προχώρησαν το θέμα, κάτι το οποίο το χαιρετίζω. Χαιρετίζω επίσης και την τόλμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ακριβώ κάποια μέλη την στήριξαν. Ε, την δε προηγουμένη εβδομάδα είδαμε την απόφαση του αυτών των έξι χωρών, Ισπανία, Μάλτα, Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος, που κατά κάποιο τρόπο ανεκάλεσαν την απόφαση τους ε, για στήριξη, εκ μέρους των στήριξη της Κομισιόν. Όμως, από ό,τι έχω καταλάβει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το ότι κάποια κράτη-μέλη ανακάλεσαν μπορεί να εμείνει στην πρότασή της. Και από ό,τι ξέρω, ε, είχατε κάνει κάποια εξόλωση των πραγμάτων, ήταν πάρα πολύ ορθή. Τότε λοιπόν σας είχαν στηρίξει τα κράτη-μέλη, αν όχι όλα. Αν και όχι όλα τότε, μάλλον. Άρα για πέστε μας τότε, τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε. Τρίτον, τον Νοέμβριο έχουμε την ε, Σάντσε Τσικάντ στην Βραζιλία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε εκεί να παραστούμε και να κατεβάσουμε κάποια πρόταση όπως και πέρσι, δηλαδή το να έχουμε κάποιες ε, πληροφορίες, κάποιες εκθέσεις όσον αφορά τις ελεγκτικές δραστηριότητες ε, της ΙΚΑΝΤ. Επομένω, να έχουμε αυτά τα δεδομένα, αυτέ τι πληροφορίε που θέλουμε, τόσο να μπορέσουμε να προπαρασκευαστούμε για την Ικάντου του Νοεμβρίου. Κάτι άλλο επίση, από πλευρά ειδικού βάρου αυτών των αναλύσεων, κύρου του. Εγώ νομίζω ότι έχει προσωρινό χαρακτήρα αυτή η απόφαση των κυβερνήσεων αλλά και η πρόταση της Κομισιόν και βασίζεται στο ότι υπάρχει πρόθεση να βρεθούν κάποιες ε, μελέτες επιστημονικέ σε σχέση με, το, με, με την κατάσταση των ελευθερικών πόρων για τον κόκκινο τόνο και να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Είναι ακριβής ή όχι η εντύπωση που έχουμε τώρα. Τέλος πάντων, ε, θέλω να σας πω ότι προβληματιζόμαστε, ανησυχούμε γιατί δεν... Να, να, να, να δούμε ε, το πώς θα καταλήξουμε στο ιστολογικό. Δηλαδή, να τεκμηριώσει μια πολιτική απόφαση η επιστημονική μελέτη και να μην έχουμε το ανάποδο. Υπάρχει πρόβλημα με τους ελευτικούς πόρους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά και με ανησυχεί, με φοβίζει. Και σας το λέω μα, ότι έτσι όπως τώρα έχει η πολιτική συγκυρία, ότι θα υπάρχει μια τάση κάποιες επιστημονικές μελέτες να αλλάξουν κάπως τη, την αρχική εντύπωση, την αρχική πρόθεση. Κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, σας λέω, υπάρχει αυτό το ρίσκο και σας το επισημαίνω εν ώψη της ε, επερχόμενης Κύριε Στίβενσον, έχετε το λόγο. Στίβενσον. Έχουμε προϊστορία θλιβερή όσον αφορά την έλλειψη πυγμής εκ μέρους του Συμβουλίου, έλλειψη συνέπειας εκ μέρους της ΕΚΑΔ, όσον αφορά τους αλληλευτικούς πόρους. Εγώ συμφώνησα μετά όσο αποφασίστηκα στο Μόνακο. Ε, γι' αυτό το έκανα γιατί θέλω να υπάρχει ένα καμπανάκι ούτω ώστε να ξυπνήσει, να, να δραστηριοποιηθεί η ΚΑΤ. Να ξυπνήσει στη συνάντηση του Νοεμβρίου και κάτι επιτέλους να κάνει. Οπότε, να δούμε τι θα κάνουμε με, τα, με, τους, με τον ξηφία. Γιατί με τον ξηφία υπάρχουν κάποια λεφτική πορεία επαρκής, ας πούμε, στις Αζόρες. Και αν πάει κανένα και δει αυτό το παράδειγμα του ε, όσον αφορά τον ε, τόνο Bluefin, ίσως καταλήξουμε, παρά το ότι υπάρχει κάποια παριά των πόρων, να μην μπορεί κανένας ποτέ να πουλήσει το, το, το, την ψαριά του. Το αλλιεύουμε επομένω, ε, τώρα ακούσαμε τι είπατε και ο κ. Ρομέρο τι είπε, θα μας εκπροσωπήσετε, θα, θα προβάλλετε τις ε, απόψεις μας με πυγμή και άρα θα πει κανείς που στην τώρα διάσωση των αλληλευτικών πόρων στην Βραζιλία ή όταν έρθει η τωρα η ποτε η λαμβανεται καποια μετρα τωρα διασωση των αλληλευτικων πορων στην βραζιλια η οταν ερθει η ωρα της Ντόχα τότε τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Άρα θα να μην το ξεχνάτε κύριε Πρόεδρε εσείς και ο κύριος Ζωμέβα τον θα να μας εκπροσωπήσετε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Να σας πω και εγώ τώρα δύο λόγια. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ακούσω την γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά από τη Γενική Διεύθυνση Αλληλείας για αυτός που μίλησε προέρχεται από το περιβάλλον και άλλωστε είναι σαφής η προστριβή, η σύγκρουση που έγινε μεταξύ αυτών των δύο διευθύνσεων της Κομισιόν. Καταρχήν επομένω το πάνω χέρι το είχε το περιβάλλον. Σε δεύτερη φάση όμως θα κατησχίσουν τα επιχειρήματα της ε, Με Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ρωμέβα, οι υπουργοί θα κρίνουν και τελικά πάνω χέρι το έχει το περιβάλλον. Έχουμε αυτό το ψήφισμα τη 9 Σεπτεμβρίου ή όποτε είναι. Έχουμε την απόφαση τη 21 η Σεπτεμβρίου των κρατών μελών όπου είπαν τα κρατημέλη δεν θέλουν να στηρίξουν αυτή την πρόταση. Όμως θα γίνει σαν τη ΣΥΤΙΣΙΚΑΤ και να δούμε αν θα πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Συγγνώμη, αλλά εδώ υπάρχει κάποιο είδου ε, χάος, δηλαδή τι θα προβάλλετε και την πρότασή σα την πρόταση των κρατών μελών, τι θα κάνετε στην ΕΚΑΤ, μα έχετε μπερδέψει. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις τελικά τι θέση θα έχει η Ένωση των κρατών μελών. Ποιο θα πάει εκεί πέρα από πλευρά Κομισιόν, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο ή Αλία. Και φαντάζομαι ότι το σχέδιο ανάκτησης πρόκειται να αναθεωρηθεί. Θα μπει ο κοινός τόνος στο πρώτο παράδειγμα ΣΥΤΕΣ, θα έχουμε κάποια περιοριστικά μέτρα, θα έχουμε το σχέδιο ανάκαμψης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα αποφασίσει σχετικά στα περιθώρια των αποφάσεων της ΙΚΑΔ. Όμως, φανταζόμαστε ότι θα υπάρξουν τέτοια περιοριστικά μέτρα και σχεδίο ανάκαμψης. Τελευταίο θέμα τώρα. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι ε, σχετικό κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, αλλά, αλλά όταν οι ΣΥΤΕΣ στα παραρτήματα, εντάσσει κάποια ψάρια, κάποιου ελευθερικού πόρου, διαβουλεύεται, συμβουλεύεται σε σχέση με την ΦΑΟ κάποιου ειδικού. Και εκείνοι αξιολογούν το τι θα γίνει στην ΣΥΤΕΣ με τα σχετικά ψάρια. Για πετε μας επομένω, αυτή η εκτίμηση πλευρά ΦΑΟ προς ΣΥΤΕΣ Πότε θα γίνει, νομίζω ότι υπάρχει πάντως κάποιο χρονικό όριο που είναι 24η Οκτωβρίου. Θα γίνει επομένω μια τέτοια συνάντηση, μια τέτοια συνεδρίαση των εμπειρογνωμόνων. Οι επιστήμονε είναι εκεί πέρα, αλλά συνήθω ε, λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τη των πόρων παρά το περιβάλλον. και τη σχέση εμπορίου και αληθική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτέ οι ερωτήσει αφορούν και την αλληλεγγύη και το περιβάλλον. Εσεί απαντήστε με όποια σειρά θέλετε. Αλλά μην μιλάμε μόνο το περιβάλλον, στην Επιτροπή Αλληλεία είμαστε. Ε, Θέλει κάποιο από τη διεύθυνση τη ε, Έχετε το λόγο. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να μην σχολιάσω περί διαφορετικών ε, απόψεων σε επίπεδο επιτροπών της ε, υπηρεσιών της Επιτροπής. Η πρόταση είναι πρόταση της Επιτροπής, την έχουμε υιοθετήσει όλοι δηλαδή από κοινού και περιλαμβάνει την υποβολή για τα κράτη-μέλη μίας προσωρινής ε, ταξινόμησης υπό τον τίτλο Α που δεν απεδέχθησαν τα κράτη-μέλη και σε τούτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει, δεν έχει υποστηριχθεί η πρόταση του Μοναχικού πλην όμως, όπως είπε και από το περιβάλλον, την τελική απόφαση δεν την έχουμε ακόμη κρίνει, δεν έχει κρυθεί το ζήτημα εν τέλει και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το Μάρτιο να έχει καταλήξει για τη συνεδρία του Μαρτίου και στην απόφασή της να λάβει υπόψη και τα συμπεράσματα της συνεδρίας του ΚΑΤ και τα νέα επιστημονικά στοιχεία που θα έχουν ενδεχομένως στη διάθεσή μας μέχρι τότε για την ε, περιγραφή της ε, κατάστασης ε, της σχετικής με τον ερυθρό τόνο και τα μέτρα για την προστασία του είδους αυτού. Φρονώ ότι είναι μεγάλη αδικία να ισχυρίζεται κανείς ότι τίποτε δεν έχει γίνει, ότι δεν έχει αναλυθεί καμία πρωτοβουλία. Υπάρχει μέτρα προστασία εδώ και τρία χρόνια, ένα πρόγραμμα για την προστασία του ερυθρόπτερου πτώνου ε, πρόγραμμα προστασίας το οποίο όμοιο του δεν έχει στον κόσμο, σημειώνω. Είναι το πληρέστερο πρόγραμμα με στόχο την, ε, τον έλεγχο, την ανάπτυξη του ελέγχου αυτής, αυτού του είδους της αλίας και τα κράτη-μέλη έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να ελέγξουν την αλία και εμείς το ίδιο προσπαθούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη ε, τα οποία πολλές φορές ειδικά τα άμεσα εμπλεκόμενα έχουν επιδείξει και πολύ μεγάλη πολιτική παρησία στον έλεγχο του στόλου, την ε, διάλυση πλοίων ή την ε, αγκυροβόληση πλοίων κατά την διάρκεια τις ε, αλλιευτικές περιόδου και τα νέα μηνύματα που έχουμε από τη φετινή ε, περίοδο παραμένουν πολύ αισιόδοξα, πολλά υποσχόμενα και πολύ φορές να μιλήσουμε με το, με το Κοινοβούλιο για ε, περισσότερες λεπτομέρειες, ας σας ενδιαφέρουν. Για το ΕΛΚΑΤ είναι ίσως πρόημο να εκφράζει κανείς ανησυχίες, ούτως ή άλλως θα προηγηθούν πολλές συζητήσεις με πολλούς από τους εμπλεκόμενους παράγοντες και η Επιτροπή την απόφασή της θα τη λάβει με ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις και στο επιστημονικό πεδίο. Πάντως σημειώνω αμέσως ότι δεν προβλέπεται να γίνει αξιολόγηση αποθεμάτων εφέτος. Και μάλλον θα ε, ανανεωθεί ή θα ε, συμπληρωθεί με πιο επίκαιρα στοιχεία η περσινή έκθεση του ΕΚΑΠ ε, στην προσοχή του συνεδρίαση, στην προσοχή συνεδρίαση του Συμβουλίου αυτού. Σημειώνω δε ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για μορατόριου, για διακοπή δηλαδή αλίας στην προηγούμενη έκθεση. Εξετάστηκε το ενδεχόμενο του μορατόριου, αλλά δεν υιοθετήθηκε η πρόταση αυτή στην τελευταία συνεδρίαση. Αυτά λοιπόν και εμείς βεβαίως ενθαρρύνουμε τους επιστήμονες ε, να ε, ασχοληθούν με το θέμα αυτό στην προσοχή τους ε, συνεδρίου στο δυνατό, να εξετάσουν τα κριτήρια και βεβαίως ανάλογα τις αποφάσεις τους ε, περί τοποθέτησης προς τα κριτήρια τις λαμβάνουν και με βάση δεοντολογικά ε, δεοντολογικές αρχές, ηθικό γνώμονα δηλαδή, αν πρέπει να παρέμβουν σε θέματα που ανήκουν προς το πεδίο της ΙΤΕΣ. Και πάντως ασφαλώς θα πρέπει εκείνοι που είναι οι ειδικοί για τον ερυθρό τόνο και δεν είναι και τόσο πολύ αυτοί, θα πρέπει πιστεύουμε να συμμετάσχουν στις σχετικές εργασίες, διότι εκεί θα μελετηθεί ακριβώς η κατάσταση του είδους, τα αποθέματα δηλαδή, ε, βιολογική μελέτη των αποθεμάτων του είδους. Ασφαλώς η ΣΥΤΑΣ αποδίδει μεγάλη σημασία στο είδος αυτό, Ασφαλώς είναι σαφές το πολιτικό μήνυμα της πολιτικής σημασία που αποδίδεται, σαφώς το έχουν αντιληφθεί οι ηγέτες οι Ευρωπαίοι το μήνυμα αυτό. Απλώς θα ήθελα για σας να σημειώσω ότι είμαστε στο πλαίσιο πολυμερών διαπραγματεύσεων με πολλούς άλλους παράγοντες, φορείς και η ΑΛΙΚΑΤ. Ανεξαρτήτως της θέσεως που θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει απόρριψη από άλλα κράτη-μέλη μια τέτοια πρόταση, είτε για μορατόριο από την Αλικάτ, είτε στο πλαίσιο του ΣΥΤΕΣ, ε, εγγραφή στο πρώτο παράρτημα. Με ό,τι συνέπεια μπορεί αυτό να ε, επιφέρει ως προς την κατάσταση του είδους, ως προς το είδος του τόνου, πράγμα στο οποίο δεν θα επεκταθώ τώρα, δεν είμαι σε θέση να το πράξω αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι εμείς προσφέρουμε στην Αλικάτα, εγγράφοντας τον, στο, εγγράφοντας το πρώτο παράρτημα, υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσει μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα, να στραφεί δηλαδή κατά, να γυρίσει μπούμεραν και για τον κόκκινο, τον ερθρό τόνο στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε όμως τώρα και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιβάλλοντος τη ε, Γενική Διεθνή των Περιβάλλοντων από την Επιτροπή. Ναι, ευχαριστώ. Αν επιτρέπετε, θα ήθελα να πατήσω σε κάποια εναπομείναντα ερωτήματα, γιατί δεν καλύφθηκαν όλα από τον συνάδελφο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα σχετικά με τι ε, διαδικασίε. Και θα επισέλθω σε κάποιες λεπτομέρειες. Όπως είπα και νωρίτερα, η απόφαση λαμβάνεται σε δύο βήματα. Τώρα έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο βήμα, δηλαδή το αν θα μπορούσαμε να ε, χρηματοδοτήσουμε την πρόταση. Η απάντηση είναι ότι δεν είμαστε σε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε μια τέτοια πρόταση. Μια τέτοια απόφαση όμως δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι αποκλείεται στο μέλλον να προσφερθεί υποστήριξη κάποιας άλλης πρότασης που θα υποβληθεί στις 14 Οκτωβρίου από τα όργανα του ΣΥΤΕΣ. Ως προς τη θέση και εδώ έχουμε να κάνουμε μια ε, σταθερή πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ε, στην κοινή θέση μιλάμε όλοι με μία φωνή. Η ΣΥΤΕΣ καταθέτει μία πρόταση για απόφαση Συμβουλίου. Μία πρόταση η οποία θα ε, προχωρήσει προς έγκριση στα τέλη Δεκεμβρίου αρχικά Ιανουαρίου. Η πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου συζητείται πρώτα στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και στη συνέχεια υιοθετείται από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος με ειδική πλειοψηφία και την απόφαση τη λαμβάνει το Συμβούλιο για όλα τα διαφορετικά θέματα που θα συζητήσει το ΣΥΤΕΣ 15. Υπάρχει λοιπόν ε, εξέλιξη και σε αυτό και σε άλλα θέματα. Και θα υπάρξει και η δυνατότητα. Εσεί υπενήχθηκατε ότι είναι αργά πια. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Υπάρχει ακόμη ευκαιρία και εμεί είμαστε στρατευμένοι σε αυτήν την υπόθεση και θα επανέλθουμε στα τέλη του τρέχοντος στι αρχέ του επόμενου έτου. Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΣΥΤΕΣ απαρτίζεται από τις διαχειριστικέ αρχές του ΣΥΤΕΣ που, που περιλαμβάνουν εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και ασφαλώς έχουν σε αυτά τα όργανα εκπροσώπηση και τα Υπουργεία Αλίας. Η διαπόφαση λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία, πράγμα το οποίο εξηγεί γιατί δεν ελήφθη απόφαση παρά την ευρεία η υποστήριξη που προσφέρθηκε. Η πλειοψηφία δεν ήταν επαρκής, δεν ήταν ειδική δηλαδή η πλειοψηφία υπέρ τη πρώτας ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω αναφέρεται και στην έγγραφη εργασία. Για θέματα που έχουν να κάνουν ειδικά με την ΕΚΑΔ θα πρέπει νομίζω να μιλήσει ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση για τα θέματα της θαλάσσης. Ένα ιδιαίτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να απαντήσω δική σας ερώτηση, κυρία Πρόεδρε, για το εάν θα ζητηθεί γνωμοδότηση από την FAO. Κάθε πρόταση του ΣΥΤΕΣ ε, σχετική με θαλάσσια από ό,τι τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, απασχολεί ε, συνεδρίαση ομάδας εμπειρογνωμόνων, η οποία αν δεν απατώμε θα πρόκειται να συνεδρίασει το Δεκέμβριο στην FAO. Ε Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας ή μη. Ευχαριστώ να επανέλθω. Πρόεδρος. Κύριε Ρωμέα, παρακαλώ μην ε, επεκταθείτε πάρα πολύ. Πολύ σύντομα. Και για να υπενθυμίσω στον φίλο από την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡ ότι πολύ θα θέλαμε να είχαμε δεδομένα, τα δεδομένα της έκθεσης της, ε, της υπηρεσίας της αποκεντρωμένης για να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι για την ΕΚΑΤ και για να μάθουμε και αν θα γίνει ε, εάν θα ληφθούν οι αποφάσεις όπως ε, θα θέλαμε και εμείς. Και για να μιλήσω τώρα αγγλικά τώρα, πρόκειται να υπαχθεί σε, στη συναπόφαση τη διαδικασία αυτή αν τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας. Κυρία Φράγκα. Να προσθέσω και εγώ μια ερώτηση πριν να απαντήσω. Το μόνο πρόβλημα με τις αποφάσεις της Επιτροπής των Επιτροπών της ΦΑΟ είναι επιστήμονες, εκπροσωπούν τα περισσότερα μέλη της ΦΑΟ. Οι δε εκθέσεις τους δεν έχουν δεσμευτική ισχύ. Είναι σαν τις που μας δίνουν και εμάς. Συμβουλευτικές. Για πέστε μας εσείς του περιβάλλοντος. Πάρα πολύ πολύ αυτή η πρόταση, ούτως ώστε να πάει στο πρώτο παράρτημα ο κόκκινος τόνος. Ε, θα βάλετε και άλλα είδη ή μόνο τον κόκκινο τόνο ή στο πρώτο παράρτημα. Άλλα είδη, ε, ακόμα και φυτικά, τα οποία είναι υπό διακινδύνευση. Σε διακινδύνευση μάλλον. Μας τα πει αυτά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, παρακαλώ, και να κλείσουμε με αυτό το τις διάταξεις. Um, maybe to start with your first question. In ναι, για να ξεκινήσω με την πρώτη σας ε, ερώτηση. Στο έγγραφο εργασίας θα δείτε ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως ε, τα, κίνησε πιο πολύ τον ενδιαφέρον, το, να, το είδος ε, του ερυθρού τόνου, του αθλατικού. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε και με έναν κατάλογο διαφορετικών προτάσεων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται διάφορα είδη ε, θαλάσσια, προτάσεις που έχει δει η Διαχειριστική Επιτροπή για διάφορα είδη ε, ηχθείων που υπάγονται στο δεύτερο παράρτημα. Και επίσης πρόταση για ερυθρά και ρόδαλη γαρίδα που ε, δεν καλύπτονται στο δεύτερο παράδειγμα. Αυτά. Νομίζω ότι μπορείτε να τα δείτε στα συμπεράσματα της ε, συνεδρίασης. Για το ερώτημα το σχετικό με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου θα σήμαινε η υπαγωγή στο άρθρο 322 της Νέας Συνθήκης, Συνθήκης Λισαβόνας δηλαδή, που δεν προβλέπει προς το παρόν διαδικασία συναπόφασης. Ούτε στην τωρινή, ούτε στην συνθήκη της Λισαβόνου. Ούτε στην Νίκαια, ούτε στην συνθήκη της Λισαβόνου. Δεν ισχύει λοιπόν η διαδικασία αυτή. Ποιο είναι το πρόβλημα. Η έκθεση της ελεκτικής αρχής. Φαντάζομαι ότι θέλετε να μας διαβάσετε το νότερο δυνατό. Τι λέει η Κομισιόν. Πρόεδρε, ασφαλώς θα χρειαστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Αλλά επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να επαληθεύσω. Σήμερα ή αύριο θα σας απαντήσω πάντως. Ωραία, καλά, τότε θα, κάν θα, θα περιμένουμε την Κομισιόν και θα το μελετήσουμε. Ευχαριστούμε και τη Γενική Διεύθυνση του Περιβάλλοντος δεν θέλω να αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ παρά να μεροληπτήσω υπέρ τη διεύθυνση Ελία, μια και είμαστε εδώ η Επιτροπή Ελία. Και έτσι ολοκληρώθηκε η ημερησία διάταξη και περνάμε στο επόμενο σημείο του υπαριθμών 12 που είπαμε ότι θα αφορά την καταπολέμηση τη πειρατεία και έχουμε ένα σχέδιο κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά ε, τις, τι τις προτάσεις και συστάσεις που έχουν διατυπωθεί ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η πειρατεία στον Ινδικό. Ποιος είναι εδώ? Ο κύριος Μάλετ. Έχετε το λόγο. Ελάτε, ελάτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που συμπεριέλαβε το θέμα αυτό στην ημερήσια της διάταξη για σήμερα διότι για κάποιους λόγους αυτό το σχέδιο νομοθεσίας ε, πέρασε από το δίχτυ ε, και δεν είχε εντοπιστεί ως νομοθετικό θέμα το οποίο θα έπρεπε να παρακολουθηθεί από την Επιτροπή Αλληλείας ε, του Κοινοβουλίου. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο λοιπόν το να μπορέσουμε να κάνουμε μια πρώτη παρουσίαση αυτής της νομοθετικής πρότασης για... προς τα μέλη της Επιτροπής. Καταρχήν, δύο λόγια για το τι ακριβώς συζητάμε. Πρόκειται για μια πρόταση για ένα κανονισμό πλαίσιο που θα μετατρέψει σε κοινοτική νομοθεσία μια σειρά συστάσεων της Γενικής Επιτροπής Αλληλείας για την Μεσόγειο. Είναι πιθανόν ε, κάποια από τα μέλη της Επιτροπής να μην γνωρίζουν τις εργασίες της Επιτροπής αυτής. Αλλά πρόκειται για τον διαχειριστικό οργανισμό ο οποίος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των ε, ενδιάμεσων υδάτων. Είναι ένα μεγάλο τομέα λοιπόν που καλύπτεται από αυτήν την, επιτροπή, την Γενική Επιτροπή Ελληνία για την Μεσόγειο. Υπάρχουν εννέα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα που είναι μέλος αυτής της Επιτροπής και συμμετέχουν στις ετήσιες συνεδριάσεις τη Επιτροπής αυτή. Ο λόγος για τον οποίο τώρα προτείνουμε κανονισμό είναι ότι στο παρελθόν η παράδοση ήταν να συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα τα οποία λαμβάνονταν από την Επιτροπή για τη Μεσόγειο στα ανετήσιο κανονισμό για τα ΤΑΚ και τις ποσοστώσεις ήταν μία από τις πολλαπλές προσωπιστήκες που μπορεί κανείς να βρει σε εκείνες τις ε, κανονισμούς. Ε, φέτος όμως ε, στην ε, Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ θεωρήθηκε ότι ήταν πιο σκόπιμο εν ώψη της Λισαβόνας και της μεγαλύτερης διαφάνειας να πάρουμε τις διατάξεις που υιοθέτησε η GFCM και να τις τοποθετήσουμε σε τρεις μόνιμους κανονισμούς που θα αποτελέσουν ένα πλαίσιο που με τη σειρά του θα μπορεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις συστάσεις που θα υιοθετούνται από την GFCM. Διατάξεις δηλαδή για μέτρα διαχείρισης των αλλιευμάτων στη συγκεκριμένη ρυθμιστική περιοχή. Επίσης να καταστήσω σαφές στην Επιτροπή ότι οι συστάσεις όταν υιοθετούνται ε, αποκτούν δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα συμβαλώμενα μέρη, δηλαδή τα κράτη-μέλη που είναι τα ίδια συμβαλώμενα μέρη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, μάλλον κοινότητα, έξι μήνες μετά από την υιοθέτησή τους. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, οι συστάσεις ε, της ετήσιας συνόδου του 2009 κατέστησαν δεσμευτικά, καταστέθηκαν δεσμευτικά το 2009, το Σεπτέμβριο του 2009. Ε, συντάσσονται σε δύο γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά και ε, τελευταία και στα αραβικά. Και θεωρούμε πως είναι πλεονέκτημα και γι' αυτό και οι συστάσεις αυτές, οι τμήματα αυτών κανονικά μεταγράφονταν στον κανονισμό για τα τάκ και τις ποσοστώσεις ετησίως. Υπήρχε όμως πλεονέκτημα να είναι πιο διαφανή και πιο κατανοητά στους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες όταν αυτά μεταφράζονταν στη γλώσσα τους και συμπεριλαμβάνονταν στην κοινοτική νομοθεσία. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε και αυτό που έχει υιοθετηθεί από την Κομισιόν, το σχέδιο κανονισμού, ε, στην ουσία αποτελείται από διάφορους κανονισμούς ε, συστάσεις μάλλον ε, της GFCM, της Γενικής Επιτροπής Αλληλείας για τη Μεσόγειο, που έχουν ενταχθεί και πρέπει να ενταχθούν στην κοινοτική νομοθεσία και ο τρόπος με τον οποίο προχωρήσαμε είναι να πάρουμε τις διατάξεις των συστάσεων που δεν ε, τηρούνται ακόμα, δεν καλύπτονται μάλλον ακόμα από την κοινοτική νομοθεσία. Συγκεκριμένα ένα παράδειγμα είναι ο κανονισμός για τη Μεσόγειο 1967-2006 κανονισμό που είμαι βέβαιος ότι τα παλιότερα μέλη της Επιτροπής θα τον γνωρίζουν. καθώς και ο κανονισμός 1005 του 2008 που αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2010. Έχουμε στην ουσία πάρει τις διάφορες συστάσεις της GFCM, οι οποίες είναι πλέον δεσμευτικές και τις έχουμε τοποθετήσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Και το συγκεκριμένο πλαίσιο μπορεί να αναθεωρηθεί και να τροποποιηθεί ετησίω από τη στιγμή που εκδίδονται νέε συστάσεις από την Γενική Επιτροπή Αλίας για τη Μεσόγειο. Θα μπορούσα επίσης να τονίσω ότι όπως οι περισσότερες τέτοιες ε, διατάξεις, ε, τμήμα το πιο σημαντικό τη διαδικασία δεν είναι μόνο η υιοθέτηση της δεσμευτική φύση των συστάσεων, αλλά το τι θα γίνει μετά στη συνέχεια Δηλαδή κατά την προπαρασκευαστική φάση των προτάσεων, συστάσεων που τίθεται επιτάπητος, διότι σαφώς εάν δεν προταθεί οτιδήποτε, φυσικά και τίποτα δεν πρόκειται να υιοθετηθεί. από την ετήσια συνεδρίαση. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλοι έχετε δει το σχέδιο κανονισμού, αν και υιοθετήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου από την Κομισιόν, όπως σας είπα, και αν και ήδη έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε από αυτού στο Συμβούλιο και το εξτάζουμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό λεπτομέρειες, αλλά βασικά, όπως σας είπα, πρόκειται για έναν κανονισμό που σε 31 άρθρα συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψη τις διάφορες συστάσεις που έχει υιοθετήσει η GFCM. Καταρχήν υπάρχει ένα τμήμα που ασχολείται με αυτά που αποκαλεί η GFCM περιορισμένες ε, περιοχές αλίευσης, ενώ ο κανονισμός για τη Μεσόγειο αποκαλεί προστατευόμενες περιοχές ε, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες και οι ελευτικές δραστηριότητες ρυθμίζονται και υπάρχει και ένα όργανο διαχείρισης. Έπειτα υπάρχει η χρήση των ομαδοποίητων, Μένων ε, μηχανισμών για την ε, αλίευση δελφινιών, αυτό με βάση τις συστάσεις του 2006. Έπειτα υπάρχει ένα τμήμα που αναφέρεται σε τεχνικά μέσα, μέτρα, ας πούμε τα μεγέθη των ματιών με βάση τις συστάσεις που έγιναν το 2005, 2009 και 2007 και έπειτα υπάρχει και ένα τμήμα που ε, αφορά την καταγραφή, το μητρό, τον ιολόγιο μάλλον, των εγκεκριμένων σκαφών. Είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε σαφή ιδέα για το ποια σκάφη κυκλοφορούν στο, στην περιοχή του ε, GFCM και ένα σημαντικό τμήμα είναι τα κρατικά λιμενικά μέτρα, τα οποία όπως ανέφερα και στην ε, εισαγωγή μου, πρόκειται για μέτρα τα οποία δεν, είναι, δεν υπάρχουν στους, ε, στον κανονισμό IUU, αλλά αφορούν ε, ειδικά την περιοχή της GFCM. Ορίζονται επίσης προδιαγραφές για την ανταλλαγή πληροφοριών και επίσης η παγίωση ενός πολύ, σημαντικών μηχανισμών αναφοράς για την περιοχή GFCM και που σχετίζονται τόσο με ε, την αλλιευτική προσπάθεια όσο και με τα αλλιεύματα, ε, δηλαδή αυτά που λέγονται στοιχεία task 1 και task 2, πολύ σημαντικά ώστε να τροφοδοτήσουν τη διαδικασία λήψης απόφασης στην GFCM. Και τέλος υπάρχουν και διατάξεις που αφορούν το πώς μπορεί να τροποποιηθεί ο κανονισμός από τη στιγμή που θα έχει υιοθετηθεί. Γιατί όπως σας είπα, οι συστάσεις αυτές ε, γίνονται σε αιτήσια βάση και μπορούν να ενσωματώνονται σταδιακά στον κανονισμό αυτό. Αυτή είναι η εισήγησή μου. Φοβούμαι ότι δεν γνωρίζω πώς από αυτά ήδη γνωρίζετε για την πρόταση αυτή, αλλά φυσικά είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Και η βασική μας ε, μέρημνα βεβαίως από την πλευρά της Κομισιόν είναι η διαδικασία γνωμοδότησης από την Επιτροπή σας και από το Κοινοβούλιο να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μέλετ. Όπως είπατε, πρόκειται για ένα νέο κανονισμό και υποψιάζομαι ότι δεν το γνωρίζουν πολύ καλά τα μέλη γιατί δεν ζητούν τον λόγο. Φυσικά έχουμε ορίσει εισηγητή, ε, μάλλον δεν έχουμε ακόμα ορίσει εισηγητή, θα το πράξουμε σε αυτό το χρόνο και φυσικά θα το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ε, δεν βλέπω κανένα να ζητά το λόγο. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο μας σημείο που είναι το 13, το πολιετές ε, σχέδιο για το δυτικό στόκ του Σαβριδιού του Ατλαντικού και να δώσουμε τον λόγο στον εισηγητή. Κύριε Κέλλε. Πρόεδρε, από ό,τι μαθαίνω, πρόκειται να γίνει παρουσίαση από τον ε, κύριο Ντόναχιου για τον τομέα αυτόν. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τη δική του παρουσίαση, να ακούσω τι έχει να πει, τι απόψεις έχει ενδεχομένως ε, να εκφράσει και άλλος συνάδελφος από την Επιτροπή και από εκεί και μετά θα προσπαθήσω να ενσωματώσω τις θέσεις αυτές στο βαθμό του δυνατού στην έκθεσή μου, ώστε να την έχω έτοιμη για τη μετάφραση μέχρι τα μέσα της προσεχούς εβδομάδας. Να ακούσω λοιπόν τις απόψεις των άλλων και μετά να παρουσιάσω τα συμπεράσματά μου. Η Πρόεδρος. Καλώς δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Τόναχιου, που είναι ο εκπρόσωπος του ΡΑΚ του αντίστοιχου για τα πελαγικά είδη, για τα είδη ανοιχτής θαλάσσης δηλαδή. I you for the uh, to make. Uh, ευχαριστώ. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάνω απ' όλα που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω μια σύντομη ε, πρόταση για, τον, για, το, για το σκουμπρί. Σαφρίδι λέω. Δηλαδή. για το σαφρίδι. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν στη διαχείριση στις ε, πρωτοβουλίες ε, του Ράκανικ της θαλάσσης και τις προτάσεις για ενσωμάτωση στο κείμενο. Και εν τέλει κάποια σχόλια μόνο για την όλη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο ε, η οργάνωσή μας ε, εξετάζει αυτά, αυτές τις προτάσεις. Πριν περάσω λοιπόν σε λεπτομέρειες, ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το να δούμε εδώ πέρα ότι έχει πολύ μεγάλη ε, κατανομή, πολύ μεγάλη διάχυση αυτό το απόθεμα ε, του Σαφριδίου από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τη Δυτική Αχθή Ακτή της Ιρλανδίας, το Βυσκαϊκό Κόλπο και ε, ακόμη και με κομμάτια της ε, μάχης το σαβρίδι είναι ένα είδος το οποίο βρίσκεται περίπου στα μισά υψομετρικά των ε, υδάτων και ε, αλλιεύεται με ε, τράτες ανοιχτής θαλάσσης. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ εδώ στην οικονομική αξία της ε, προσπάθειας μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αλίευμα 120.000 τόνων το χρόνο, με, πρώτη, με αξία πρώτης πόλης 35 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 10 με 20% του ετήσιου εισοδήματος ως προς την αλίευση ανοιχτής θαλάσσης για ορισμένους. Έχουμε απασχόληση περίπου 6.000 εργαζομένων και 637 σκαφών. Από την πιο περιορισμένη, αν θέλετε, περιοχή της ε, ε, του Βυσκαϊκού μέχρι την πιο πλούσια περιοχή της Δυτικής Ιρλανδίας και της Βόρειας Θάλασσας. Εδώ θα ήθελα να να δώσω κάποιες πληροφορίες υποβάθρου, γενικές πληροφορίες προς ενημέρωση. Μέχρι το 2003 είχαμε την ε, αναλυτική αξιολόγηση και τις συμβουλές που έφερε για τα θέματα αυτά. Πλην όμως, ε, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα ως προς την ε, αξιολόγηση και ως προς τη συμπεριφορά του αποθέματος και η αναλυτική αξιολόγηση αποσύρθηκε στην, ε, το, μετά το 2006, τρία συγγνώμη, τελευταία δηλαδή ήταν το 2004. Και επίσης είχαμε μεγάλο πρόβλημα σε κάθε Συμβούλιο Αλίας από τις προτάσεις που παγίως υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειωθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο αλίευμα, ενώ αντίστροφα εμείς προτείναμε να διατηρηθεί στο, ε, στο του, στα τωρινά του επίπεδα. Επίσης, δεν ξέραμε εάν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ 30 και 40% παρουσιάζοντας τα αποθέματα μεταξύ διαφορών ετών. Προφανώς δεν υπήρχε ε, σχεδιασμός μακροχρόν, μακροπρόθεσμος και ως εκ τούτου θα έπρεπε ε, να αναζητήσουμε μία πρωτοβουλία σε σχέση με το θέμα αυτό και είπαμε ότι θα πρέπει να, να γνωριστεί ότι υπάρχει πρόβλημα προς την ε, επιστημονική αξιολόγηση και έτσι ε, ειδικοί ερευνητές εκλήθησαν ε, να μας προσφέρουν κάποιες ιδέες. Και έτσι θεσπίστηκε μια ομάδα μελέτης, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και είναι ενδιαφέρον ότι όταν υπάρχει πραγματικός διάλογος και πραγματική κατανόηση μπορούμε να βρούμε λύσεις. Και οι επιστήμονες είπαν ότι θα προσπαθήσουν να βρουν ε, λύσεις για την διαχείριση των υποθεμάτων μακροπρόθεσμα με αποτέλεσμα στην ομάδα αυτή εστίασης Focus Group να υποβληθούν προτάσεις ε, αρκετά πρωτότυπες, αρκετά αποτελεσματικές κιόλας για την ε, διαχείριση των αποθεμάτων. Αυτή η νέα λοιπόν πρωτοβουλία, στην οποία δεν θέλω να αναφερθώ λεπτομεριακά και κυρίως δεν θέλω να φέρω τις ε, τα οικονομικά, μάλλον τα, τους, τους μαθηματικούς τύπους με βάση τους οποίους ε, εξετάζουμε τα θέματα αυτά, ε, διαπιστώνει ότι δεν είχαμε πρόβλημα μόνο ως προς την ε, συλλογή των δεδομένων, και είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τριετή υπολογισμό σχετικό με το Σαβρίδι και με κανόνα ως προς την ε, συγκομιδή, ως προς την παραγωγή ο οποίος θα ίσχυε για ένα μέρος των ΤΑΚ και το υπόλοιπο θα κάλυπτε. Μία περίοδο εννέα έτη. Φυσικά εδώ πέρα δεν βλέπετε τα στοιχεία τα οποία έχω να σας παρουσιάσω διεξοδικά, αλλά δίνουν μια κάποια εικόνα θα έλεγα. Και εν τέλει βλέπουμε ότι αυτή η μικρή ομάδα εστίασης προτείνει στους επιστήμονες ε, λύσεις ε, που εξασφαλίζουν και τη βιωσιμότητα του αποθέματος και βέβαια σταθερότητα για τον κλάδο τον ίδιο και βέβαια προστασία των συμφερόντων των εμπλεκομένων. Έχουμε λοιπόν διάφορους τρόπους εμείς από το Pelagic Crack να εξετάζουμε τα θέματα αυτά. Έχουμε δει και συζητήσει με την ε, Εκτελεστική Επιτροπή και έτσι τον Ιούλιο του 2007 κάναμε αυτές τις προτάσεις. Και από την άποψή μας ε, κληθήκαμε να ε, ζητήσουμε από τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα να αξιολογήσει το έργο μας, πράγμα το οποίο έγινε και μάλιστα έγινε αποδεκτό ε, αυτό το οποίο προτείναμε εμείς ως μια συνετή πρόταση για την προστασία του είδους. Τα τάκ λοιπόν τα οποία είχαν οριστεί για το 2008 και το 2009 για τον ε, για το Σαβρίδι είχαν ε, βασιστεί σε αυτά τα σχέδια του ΡΑΚ. Και έτσι ερχόμαστε στην πρόταση της Επιτροπής φέτος, τον Απρίλιο, όπου είδαμε μία σειρά συνεδριάσεων στο Πελάτς Κράκ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και μία σύσταση τον Ιούλιο, που υποβλήθηκε τον Ιούλιο σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, δεν θέλω να πω ότι έχοντα εξετάσει και τα θέματα αυτά σε λεπτομέρεια με τον πρόσωπο τη Επιτροπή, θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι σύμφωνα με τι προτάσει του Pelagic Crack. Πλην όμως υπάρχουν δύο προτάσεις, τις οποίες θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και χρειάζονται δύο τροποποιήσεις για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε ορισμένα πράγματα. Και για να σας δώσω σύντομα κάποιες εξηγήσεις. Το άρθρο 6.2 ασχολείται με το παραλίευμα. Ε, πράγμα το οποίο εμάς δεν μας απασχολεί ε, ειδικά γιατί είναι ενσωματωμένο μέσα στο σχέδιο και μιλούμε για περιπτώσεις κατά τις οποίες το Σώμα των Επιστημών δεν είναι σε θέση να υπολογίσει το παραλίευμα μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονιά, μέσα σε ένα δωδεκάμινο. Εδώ έχουμε το μέγιστο ποσό των τελευταίων 15 ετών, που δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 5% σερολογία και λέμε ότι ούτε λογικό είναι, ούτε δίκαιο να επιβάλλεται ένα τέτοιο όριο. Θα σε εξηγήσουμε γιατί. Και επίσης θεωρούμε ότι επιβάλλει υπερβολικό κόστος ε, προβλήματα στους, ε, στον κλάδο, ε, δηλαδή τους επιβάλλει κόστος το οποίο δεν υπάρχει λόγος να αναλάβουν. Αν δείτε λοιπόν στον ε, κατάλογο που έχουμε παρουσία, να παρουσιάσουμε εδώ, το 1996 τα ποσοστά ε, των ε, παραλίευμάτων ήταν πάρα πολύ ψηλά. Είχαμε 4% των συνολικών αλλιευμάτων. Αλλά τα τελευταία 15 χρόνια σε μέσο όρο έχουμε μόνο 0,8% επί των συνολικών ε, αλλιευμάτων ως αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν το 1996, το οποίο δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικό έτος, να περιληφθεί σε αυτόν τον υπολογισμό. Και πέραν αυτού, η Επιτροπή δεν προτείνει 4%, αλλά 5%. Εάν δεν είναι σε θέση να υπολογίσει παραλίευματα, παραπίπτοντα αλίευματα. Όχι, ε, θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί τόσο υψηλό ποσοστό για ένα έτος στο οποίο δεν υπάρχει σαφής εικόνα ε, με την οποία μπορούν να υπολογιστούν τα παρέμπιπτου αλλιεύματα και ελπίζω να με κατανοείτε σε αυτό που θέλω να πω. Για τα παρεμπίπτοντα λεύματα λοιπόν λέμε, εμείς προτείνουμε ένα διαφορετικό τρόπο υπολογισμού με ε, αναφορά στα, τελευταία 15 ετία και τα σχετικά παραλιεύματα. Και αν τύχει, πράγμα το οποίο δεν περιμένουμε να συμβεί βέβαια, αλλά αν τυχόν τύχει να μην μπορούμε να υπολογίσουμε παραλιεύματα, θα παίρνουμε μέσω όρο των τελευταίων 15 ετών. Πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι και λογικό και δίκαιο δεδομένων των στοιχείων που σας παρουσιάζουν. Τελευταίο στοιχείο. και διαφωνία που έχουμε είναι αυτή με, η σχετική με το άρθρο 11.2. Είναι η δυνατότητα πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές. Ίσως λοιπόν θα πρέπει εδώ να εξετάσουμε και πάλι τον πίνακα που είχα παρουσιάσει στην αρχή ως προς, τον, ε, ως προς την κατανομή του είδους αν δει κανεί λοιπόν την, τον χάρτη στη Βόρεια Θάλασσα, το 4Β, τον οποίο φυσικά οι ερμηνεί δεν βλέπουν, δεν μπορεί να βγει το αλίευμα αυτό ούτε στα, στις νήσους Σέτλαντ, ούτε στην Ορβηγία, εάν γίνει εκεί η αλίευση. Και αν τυχόν αλλιεύει κανείς στο 7D, στη μάχη δηλαδή, με σημαντικά αποθέματα εκεί Ζαβριδίου, ε, πάλι δεν μπορεί κανείς να πάει με βάση την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ε, Δυτική Ιρλανδία, με βάση πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά η κατάσταση δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει. Ξέρουμε ότι αυτό το έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θεωρούμε ότι δεν μπορεί να παραμένει το πρόβλημα αυτό. Είναι υπερβολικά δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εμείς Έχουμε εδώ να κάνουμε και με ζητήματα ελέγχου και προτείνουμε να αναθεωρηθεί η σχετική πρόταση και πιστεύουμε ότι είναι ευχερής ε, η αναθεώρηση Τη σχετική διάταξη εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του κανονισμού 805 του 98 που αφορά τις, ε, τον εξοπλισμό που χρειάζεται να έχει ένα σκάφος για να εκφορτώσει το αλίευμά του σε συγκεκριμένη περιοχή. Αυτές είναι οι δύο διαφωνίες μας. Κατά τα άλλα, μας ικανοποιεί το γεγονός ότι αντικατοπτρίζονται οι ε, λεπτομέρειες των προτάσεών μας και τα ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν ε, κατά τρόπο ικανοποιητικό. Τώρα θέλω να αναφερθώ εν συντομία σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης για το Σαβρίδι. Ίσως δεν είστε νήμεροι, αλλά πάντως ε, οι προτάσεις αυτές αποδεικνύουν την ε, σημασία των διαχειριστικών ε, συμβουλίων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα ΤΑΚ αποδεικνύεται ήταν πολύ χρήσιμα και ασφαλώς και εσείς θα είσαστε ικανοποιημένοι. Εδώ έχουμε μια πολύ καλή περίπτωση προσέγγισης από την βάση και όχι επιβολής άνωθεν επιλογών όπως έχουμε δει στο παρελθόν ε, στην Αλία, πράγμα το οποίο οφείλεται σε μια καλή εταιρική σχέση, συνεργασία μεταξύ του κλάδου και του, του επαγγελματικού κλάδου της Αλίας δηλαδή και του επιστημονικού κλάδου. Και έτσι είναι δυνατόν ε, να αντιμετωπιστούν υφιστάμενα προβλήματα και να προβλεφθούν ενδεχόμενα μελλοντικά προβλήματα. Εξασφαλίζεται επίσης η βιωσιμότητα των υποθεμάτων. Πράγμα το οποίο φυσικά μας συμφέρει όλους εμάς ιδιαίτερα στον κλάδο και ιδιαίτερα την οργάνωσή μας στην Θελάτσιο Κράκ. Επίσης αποτελεί η λύση αυτή και να παραγόντα σταθερότητα για τον κλάδο, γιατί ξέρουμε για την προσεχή τριετία που βρισκόμαστε, που, σε ποια όρια κινούμαστε με κάποια μικρές ασφαλώς διακυμάνσεις που δεν ε, διαταράσουν τις εργασίες μας. Και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει η διαδικασία αυτή πρότυπο για άλλα μακροχρόνια σχέδια διαχείρισης ε, που ενδεχομένως χωρίς να είναι απόλυτα όμοια έχουν αντίστοιχα στοιχεία, χαρακτηριστικά ή δυσκολίες. Και χωρίς ε, να θέλω να μετριάσω τους επένους ε, στο σχέδιο αυτό, μακροχρόνιο προγραμματισμό, θα ήθελα να σημειώσω και κάποιες αδυναμίες. Εμείς έχουμε αποσχοληθεί πολύ καιρό από την Πελάτσι Crack στο θέμα αυτό. Έχουμε αφιερώσει ε, πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει προγραμματισμό 18 μήνο με ε, απόφαση το 2007 ήδη και πιστεύουμε ότι πέρασε πολλής χρόνος μέχρι να έρθει τώρα, ύστερα από δύο χρόνια η ώρα να συζητηθεί το ενδεχόμενο της θέσπισης κάποιου κανονισμού. Ακόμα δεν έχει θεσπιστεί δηλαδή ο κανονισμός και γι' αυτό πιστεύω ότι χάνουμε πολύ χρόνο. Θα έπρεπε να προχωρούμε σε διαδικασίες υιοθέτησης πολύ πιο γρήγορα με μεγαλύτερη σπουδή και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε για τα τελευταία 12 λεπτά. Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας και ακριβώς όπως το γνωρίζαμε χαιρετίζουμε το ότι δείξατε ευαισθησία και ανταποκριθήκατε στις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει πάντα. Εμεί θέλουμε να διεκπαιρεώσουμε όσο γίνεται καλύτερα και πιο γρήγορα το θέμα και το, το αναθέσαμε στον επιφανή συνάδελφο κύριο, κύριο Γκάλαχερ. Διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι εδώ είμαστε συσπηρωμένοι, συμφωνούμε, τα βρίσκουμε, υποστηρίζουμε τα ΡΑΚ. Τώρα ποιος άλλος θέλει το λόγο. Κυρία Αντρές. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Εγώ θα ήθελα κάτι να ξεκαθαρίσουμε το ότι αναφέρατε επανειλημμένα το θέμα της ε, καλύτερης παραγωγής, αναβάθμισης παραγωγής, αναβάθμισης των ποσοστώσεων και ότι είναι αλήθεια ότι μιλούμε για κάποια ομάδα χωρών ε, που βρέχονται από τη Μεσόγειο και ασχολούνται με ε, αυτό που μας μιλήσατε, με το, με Σαφρίδι. Όμως αυτό δεν ε, αφορά την Ισπανία. Μιλάμε τώρα δηλαδή για το κατά πόσο αυτό γίνεται χθιάλευρα και κατά πόσο απευθύνεται στην ανθρώπινη διατροφή. Επομένω, μια που εμείς ε, εδώ πέρα διαχωριζόμαστε, παρακαλούμε να γίνει μια ειδική ρύθμιση για μας. Βιλβά. Ο επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω για τα όσα μας εξηγήθηκαν και ελπίζουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο, θα υπάρξει επίσης και ισόρροπη ε, σορβημένη άσκηση της δραστηριότητα αυτής, αλλά σε σχέση με το έγγραφο το οποίο μας μοιράσατε, θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Στο κεφάλαιο 4 ε, αναφέρεστε σε ελεγκτικά μέτρα και είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει έναν καινούργιο κανονισμό. Οπότε σας ερωτώ, τα λάβατε αυτά υπόψη. Αυτά που λέει εδώ, τα έλαβε υπόψη ο κανονισμός του Συμβουλίου ΥΟΥ Πρόκειται τα σχετικά άρθρα να τροποποιηθούν επομένω ή όχι, λαμβάνοντα υπόψη το ότι επήγει η έγκριση αυτού του νομοθετήματος και ότι επίσης τρέχουν και κάποιες προθεσμίες μέσα στις οποίες θα πρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει αυτό το καινούριο νομοθέτημα. Ε, ε, sí, eh, así el señor Turgaiz había pedido ah no perdón perdón entonces voy a pasar a dar la palabra a la señora Tanking de la Comisión Europea. Tiene usted la palabra. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Es Santa Candela, señora presidenta. Había un... <laughs> Perdone, al verla usted ya me he dado cuenta, pero aquí tenía <laughs> puesto las... Ah, Α, εκεί είσαστε. Eh, Συγγνώμη, ε, κυρία Τάγκη, περίμενα, ήρθατε εσείς, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, με μεγάλη μας χαρά να σας ακούσουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, καμία παρεξήγηση. Αυτό που θέλω καταρχήν να σας πω είναι να συγχαρώ τον ε, κύριο Ντόναχιο για τα όσα τόσο, τόσο Πλήρω μα εξέθεσε και ε, θα ήθελα να σας πω ότι δεν αφήσατε καθόλου απόψει μα. Για το δε Σαφρίδη πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία ήταν πάρα πολύ αγαστή για ε, με τα και να λάβετε υπόψη ότι όντως πιέζει να γίνει ταχεία διεκπαιρέωση κάτι το οποίο είναι δική μας ε, απόφαση επίσης. Άρα θα κινηθούμε μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ξεκινάμε πρωτοβουλία του κλάδου. Άλλωστε, όλο αυτό το θέμα. Και αυτό έχει περάσει το πνεύμα και στο Συμβούλιο, όπου η δουλειά επίσης γίνεται πάρα πολύ επικοδομητικά. Λάβαμε υπόψη αυτό που μας είπε ο κύριος Ντόναχιο, ε, και θέλω να σταθώ σε δύο σημεία που ανέδειξε κάποια προβλήματα. Αυτό έχει σχέση και με το πού έχει κολλήσει το θέμα στο Συμβούλιο. Και οι δικέ μα υπηρεσίε προσπαθούν να βρούμε κάποια λύση, κάποιο συμβιβασμό. Οπότε, θεωρούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον, θεωρούμε ότι υπάρχει εδώ συμβιβασμό όσον αφορά τον υπολογισμό του παραλιεύματος όσον αφορά την εξέβρεση κάποιων μέσων όρων και επομένως το πρότυπο το οποίο εμείς προτείνουμε είναι να χρησιμοποιηθεί το πιο υψηλό νούμερο της τελευταίας πέντα ετία. Αυτό προτείνουμε ως λύση. Τώρα όσον αφορά την διαμετακόμιση, όσον αφορά το κατά πόσο χρειάζονται κάποιε προηγούμενε συγκρίσει για το σαφρίδι και τη μεταφορά του, ε, έχουμε να προτείνουμε λύση. θα πρέπει εδώ ο συνδυασμός να καλύψει και κάποια ελεγκτικά μέτρα. Όμως να υπάρχει μία πλαισίωση νομοθετική τέτοια και μία περιγραφή του τι θα πρέπει να ισχύει όσον αφορά το χώρο αποθήκευσης του πλοίου. Έχει γίνει η αλίευση, να υπάρχουν κάποια χαρτιά έτσι να έχει γίνει λοιπόν η, κατανομή του ελεύματο και άρα μην υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τον έλεγχο εφαρμογής αυτής της ρύθμισης. Άκουσα ε, για τους ε, αγορητές που έλαβαν τον λόγο μετά την ε, εισήγηση. Άκουσα την κυρία Αντρέ, η οποία μα μίλησε για κάτι το οποίο δεν περιέχεται εδώ αλλά έχει σχέση με αυτή την πολιτική γιατί μας είπε για αναδιοργάνωση ε, των, περιοχών που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για, την, για τον υπολογισμό του ΤΑΚ. Ξέρουμε ότι εδώ πέρα είναι θέμα που και η Ισπανία και η Πορτογαλία θα ζητήσουμε κάποια λύση και θεωρούμε ότι είμαστε κοντά στην εξέβρεση της. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο σηκώνει πολύ συζήτηση, δεν μπορούμε τώρα να την κάνουμε, να πούμε τώρα στις λεπτομέρειες. Όμως, αυτές οι περιοχές που έλθουν υπόψη για να καθοριστεί το ίδιο ΤΑΚ, ελήφθησαν υπόψη πέρσι και καταλήξαν σε κάποιες προτάσεις των επιστημόνων. Προσπαθούμε τώρα να λάβουμε υπόψη τις επιστημονικές συμβουλές όσον αφορά το τι ισχύει σε κάθε ζώνη για τους αριθμού πόρους και κατόπιν να καθορίσουμε το τάκ, το μίξ του επιτρεπόμενο αλίευμα και υπάρχει το θέμα αυτό το παλιό του κατά πόσον μπορούν τα κατημέλη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους περιοχές όπου μπορούν να αλλιεύσουν Θέλουμε να υπάρχει ε, ένα σύστημα το οποίο να μην επιτρέπει να ρίχνεται κανείς ούτε να στρεβλώνεται η δραστηριότητα, ο κλάδος. Ακούσαμε την είπε και η κυρία Βιλμπά. Έχω να σας πω κυρία μου ότι η Σουηδική Προεδρία έχει σκοπό στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου να εγκρίνει έναν ελεγκτικό κανονισμό. Θα περιέχεται και ένα κεφάλαιο όσον αφορά κάποιες διατάξεις οι οποίες θα είναι εφαρμοστές όταν ισχύσει το πολιετές πρόγραμμα. Και σε αυτή την περίπτωση οι διατάξεις αυτές θα εφαρμοστούν. Και επίση θα πρέπει να έχουμε και ελεκτικέ διατάξει και στα πιο μικροπρόθεσμα προγράμματα. Πρέπει να δούμε επίση τι, ε, τι περιθώρια θα αφήσουμε όσον αφορά την ε, αποθήκευση και τη μεταφορά των, του αλλιεύματος, αλλά και όσον αφορά την εκφόρτωσή του στο λιμάνι. Ολόθερμα φυσικά και επιθυμούμε να εμφανιστεί σαν σημείο Α στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου αυτό το θέμα και νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν παράλληλα να διεκπεριωθούν αυτά τα θέματα το ένα μετά το άλλο αλλά επαναλαμβάνω στον κανονισμό αυτό θα υπάρχει ένα κεφάλαιο που θα αφορά τον έλεγχο ευχαριστώ Φράγιο εμείς ευχαριστούμε πολύ δεν ζητεί άλλο το λόγο και ο κύριος Γκάλα, κύριος ηγητής, θα λέει το λόγο για να κληρώσουμε αυτό το θέμα. Uh, ευχαριστώ, Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόναχιο που αντιπροσωπεύει το Pelagic Rack για την παρουσίασή του και για τις ε, μαθηματικές ε, εξισώσεις που μας έδειξε, τύπους που μας έδειξε. Δεν ξέρω τώρα αν τους κατάλαβαν όλοι. Πάντως ήταν σημαντικό που μας το παρουσίασε γιατί μας έδειξε με σαφή τρόπο τη σημασία και το αναφέραμε και χτες, τη σημασία της ε, συνεργασίας και ποιοι θα κερδίσουν και θα, ε, ή θα χάσουν από αυτό ο ίδιος ο τομέας της αλίας. Όχι εμείς, ούτε η Κομισιόν. Και εκείνοι αναγνωρίζουν τη σημασία της ύπαρξης ενώ μιας βιώσιμης αλίας. Πολύ σημαντική ο αλίευμα, 120.000 τόνι, ένα σωρό τομείς καλύπτονται, διάφορες μορφές απασχόλησης, 45 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, τζίρος και φυσικά αυτό πολλαπλασιάζεται γιατί αυτό είναι η χοντρική. Μιλάμε για απασχόληση πολλών ανθρώπων. Η παρουσίαση λοιπόν που έγινε σας πήρε 12 λεπτά να μας κάνετε αυτή την εισήγηση, αλλά Σίγουρα έχει πάρει ώρες και εβδομάδες και μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων και έρευνας από το Pelagic ράκ σε συνεργασία με την Κομισιόν και φυσικά έχει βρεθεί ένας καινοτόμο τρόπος για την αξιολόγηση με βάση δεδομένα και στοιχεία από τη στιγμή που υπήρξε μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και είμαι ικανοποιημένο από την τήσια έρευνα που γίνεται σε συνεργασία με την ε, Μάκρο και αυτό οδηγεί στο μαθηματικό τύπο τον οποίο έχουν ε, ξέβρει για να φτάσουν στα τάκα και στις ποσοστώσεις της αιτήσει. Πιστεύω πως εν γέννη η ανακοίνωση είναι 95% αποδεκτή Ωστόσο, νομίζω πως ε, ως αποτέλεσμα των όσων υποστήριξε ο κύριος Αντώναχιου και εξ ονόματος του Πελάζε Κράκ, σίγουρα εμένα με έπεισε ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το άρθρο 12.2 σε σχέση με την κίνηση ανάμεσα στις διάφορες περιοχές χάρτης με την κόκκινη γραμμή με έπεισε ότι δεν μπορείς όταν αλλιεύεις σε μια περιοχή 4β ή 4α ή εν πάση περιπτώσει αν δεν θυμάμαι τώρα αν είναι 6ε αν θα μπορείς ας πούμε να εκφορτώσει και να κατεργαστείς ε, το αλίευμα στην Νορβηγία ή στα Σέτλαντ, αυτό ήταν καλό παράδειγμα. Ή όταν θέλει κανεί να εκφορτώσει στην Πορτογαλία ή την Ισπανία. Εγώ θα προτείνω λοιπόν τροπολογία εδώ σε σχέση με την έγκριση και την περίμετρο που χρησιμοποιεί νομίζω η Κομισιόν. Και αυτό βέβαια σε συμφωνία με τον κανονισμό που ήδη υπάρχει. Το 850 Πιστεύω επίση ότι θα πρέπει να δούμε την ε, απαλλαγή. Είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά θα ήταν πολύ άδικο νομίζω να θα πρέπει να δούμε όχι το 96, το 16,07, Νομίζω πως δεν είναι αντιπροσωπευτικό και ορισμένες φορές χρειάζονται επεκτάσεις. Σας ευχαριστώ για αυτό και εγώ προσωπικά υποστηρίζω και την πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα να αναγνωρίσω την συνεργασία των επιστημόνων της Κομισιόν και τώρα του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες εκτίμησης. Ελπίζω πως τις επόμενες μέρες θα έχω έτοιμη την έκθεσή μου για μετάφραση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε για το Κοινοβούλιο, είτε είναι μετά τη Λισαβόνα είτε πριν, ελπίζουμε να είναι Λισαβόνα, γι' αυτό είναι η υπόθεση των Ιρλανδών, ελπίζουμε λοιπόν ότι θα γίνει αποδεκτό και από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Χωρίς να καθυστερήσω άλλο. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαδικασίες από κάτω προς τα πάνω και επικρίνω τις αναθεωρήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, αλλά αν υπάρχει μία αλλαγή που πρέπει να γίνει, θα πρέπει να είναι η θέσπιση των ΡΑΚ. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Ντόναχιο και του συναδέλφους του για την εργασία του και για την εισήγησή του και πιστεύω πως είναι φυσικά θέμα της Επιτροπής, μπορούμε να δεχτούμε το πολύ λογικό αίτημα για κάποιες ίσονο σημασία στι τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλαχερ και ευχαριστούμε και τον προσκεκλημένο μας κύριο Γκάλαχερ και την κυρία Κάνιβατ. Να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις ε, 14 ε, Νοεμβρίου και εκεί θα παρουσιαστεί και η εισήγηση του κύριου Γκάλαχερ. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ε, ακούσουμε κύριο Γκάλαχερ και ολοκληρώσαμε το 13, πάμε στο 14. Κόλπος του Βυσκαϊκού. Έχουμε και εκπροσώπους του Ωραία. Έχουμε εκπρόσωπο του Καντάβριο. Ο Γάλλος εκπρόσωπος που καλέσαμε δεν μπορούσε να έρθει γιατί είναι αλία που αφορά κυρίως στην Ισπανία και τη Γαλλία. Και θα ακούσουμε και την κυρία Αντρέση στη σεμινάρια. Για να ξεκινήσουμε, έχει το λόγο η κυρία Μπιλμπάου που είναι και η συγγετρία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους ε, του φορέα που είναι σήμερα μαζί μας. και τους ε, εκπροσώπους των αλλιέων, όπως και τους ε, επιστήμονες, το Κεωνογραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας, το Βασικό Κεωνογραφικό Ινστιτούτο για να σημειώσω και τις ε, σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί. Ευχαριστώ. Και για τις προσπάθειες που στόχο έχουν να καταστήσουν ε, βιώσιμη, βιώσιμο αυτό το Όλη αυτή λοιπόν η δουλειά καταγράφεται, είναι δουλειά που έχει να κάνει με όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πληγεί από την άσπρη από τέσσερα χρονιά της, του είδους αυτής, αυτού αλίευσης, τη διακοπή αυτού είδους αλίευσης. Εγώ ξεκίνησα εδώ και μερικού μήνε, ασχολούμαι με τα θέματα αυτά. Έχω συναντήσει εκπροσώπους του κλάδου που έχουν καταθέσει και προτάσεις για τροποποίηση. το ε, κείμενο έχουμε προβλήματα αντίστοιχα με τα παλαιότερα. Αντίστοιχα δηλαδή με αυτά που είχαμε και στο παρελθόν, έχουμε, διαφορά, έχουμε το κείμενο και έχουμε και τις προτάσεις από τον τίτλο. Το Συμβούλιο λοιπόν στα μέσα Οκτωβρίου ε, πρόκειται να υιοθετήσει νέο κανονισμό και εγώ προσπαθώ να ε, εξασφαλίσω αρκετές πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε, να κάνουμε προτάσεις συγκεκριμένε για ε, τροποποίηση των άρθρων γιατί εμεί έχουμε συνεδρία 3 και 4 ε, Οκτωβρίου, κατά τη ε, διάρκεια τη οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί η έκθεσή μου. Ε, και φάνη, φαίνεται από ό,τι μου είπα ότι πρέπει να παρουσιαστεί η έκθεση έω τι 6 Οκτωβρίου για να προλάβουμε. Άρα θα είναι ατελής η έκθεση αφού δεν θα έχουμε υπόψη τον νέο κανονισμό που πρόκειται στα μέσα Οκτωβρίου να υιοθετήσει το Συμβούλιο. Ήθελα λοιπόν να εξηγήσω ε, στους συναδέλφους αυτό το γεγονός, την κατάσταση που αντιμετωπίζω, να σημειώσω ότι θα συνεχίσω τις προσπαθίες μου μαζί με την ε, υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να ετοιμάσουμε ε, μία έκθεση με τροπολογίες λογικές, με κάποια συνοχή για να ληφθούν υπόψη βεβαίως και οι προτάσεις των συναδέλφων. Καλώς λέει η πρόεδρος, φαντάζομαι ότι θα κάνει η Επιτροπή κάποια σχόλια. Αν και δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τίποτα χωρίς πρόταση από την Επιτροπή. Παρακαλώ. Ε, καλημέρα σας. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση ότι μπορεί να εκπροσωπούμε την ε, περιοχή της Καντάμπρια, αλλά βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου. Άρα είμαι και εκπρόσωπος της σχετικής ομάδας του Συμβουλίου. Αυτά. Για να ξεκινήσω και επίσης θέλω να σημειώσω τελευταία συνεδρία στο USSR χώρα το Μάρτιο που μας πέρασε. Τον Ιούλιο δημοσιεύθηκαν τα σχόλια και έκτοτε το Συμβουλευτικό Συμβούλιο δεν έχει συνέλθει. Θα γίνει βέβαια μια συνεδρία στη Μαδρίτη και οι απόψει που σας παρουσιάζω είναι είτε του ΣΕΣΕΡ είτε προσωπικές παρατηρήσεις είτε παρατηρήσεις που ε, μου ζήτησε να υποβάλω ο κλάδος ε, της Αλίας στην Κατάμπλια. Έχουμε λοιπόν ε, εδώ και δύο χρόνια να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει βοηθήσει και επίσης μας έχουν βοηθήσει και τα τεχνολογικά Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται. Και... Έχουμε εδώ το μεγαλύτερο μέρος των ε, προτάσεων Πέντε προτάσεις. Έχω αυτές τις πέντε προτάσεις. Για αυτούς τους κανόνες εκμετάλλευσης. Έψιλον, ε, έτσι το ονομάζουμε. Αυτό θα προκύψει από το ρακ. Κάτι άλλο τώρα για το ρακ. Να υπάρχει ένα ελάχιστο τάκ. 7.000 τόνοι. Να είναι για αυτή την περιοχή αλίευσης για 20 αλλιευτικά σκάφη. Αυτό να κανονιστεί. Αλλιώς αυτό πρόκειται, οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση είναι επιζήμια για τον αλληλευτικό μας τόλο. Κάτι άλλο το, το οποίο ζητούμε είναι η περίοδος του ανοίγματο να είναι, η περίοδος του, του, του, να είναι από Ιούλιο μέχρι Ιούνιο της επόμενης χρονιά γιατί έχουμε τον ισχύοντα κανονισμό των ΤΑΚ, που είναι, που είναι ε, ΤΑΚ, ε, όρια ετήσια. Όμως, οι επιστήμονες ε, λένε ότι η περίπτωση αγοράς θα πρέπει να είναι η άνοιξη για την ε, περίοδο της αλλιεύσης. Άρα, εδώ έχουμε διαφορετική περίοδο, γιατί θα, σήμερα τους επιστήμονες θα πρέπει να φτάνει μέχρι τον Ιανουάριο ενώ έχουμε ρυθμίσει εμείς Ιούλιο με Ιούνιο. Και αυτό αποτυπώνεται και στο σχέδιο διαχείρισης. Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει η περίοδος ε, αυτή να, ε, να βασίζεται σε υπολογισμό 24.000 τόνων βιομάζας. Επίσης, έχουμε πολλούς ε, ελέγχους στο δε ε, συμβουλευτικό αυτό σώμα να έχουμε τους ελέγχους που προβλέπονται, με τους οποίους και συμφωνούμε, αν και έχουμε κάποια σημεία στα οποία διαφωνούμε ελάσσονα. Έχουμε τώρα κάποιες παρατηρήσεις που έχει υποβάλει ο κλάδος της Ισπανίας και συμφωνούν επίσης και συνάδελφοι από την Γαλλία. Πρώτα-πρώτα δεν συμφωνούμε με το άρθρο 3. Ότι δηλαδή να έχουμε τα ζώντα δολώματα και αυτό να περιέχεται στο ετήσιο τάκ, να και αυτό σαν τάκ, το δόλωμα. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδους ε, ρύθμιση στο σχέδιο πρόκειται για δραστηριότητα που έχει πάρα πολύ μικρή σημασία. Μιλάμε για 1% του αλλιεύματο. Και δεν καταλαβαίνουμε επομένω γιατί θα πρέπει να υπάρχει τέτοια ρύθμιση. Γιατί έτσι δεν θα είναι δυνατόν να ασκείται έλεγχος Δεν γίνεται, δεν, δεν, δεν μπορεί να ελέγξει κανείς πόσο έχει αλλιευθεί. Πρόκειται για πάρα πολύ μικρά ψάρια. Και γι' αυτό και εσείς ότι και οι επιπτώσεις στο συνολικό αλλιεύμα είναι αμεληταία. Τώρα σας πάω στο άρθρο υπαριθμών 13 του σχεδίου κανονισμού, εκεί όπου απαγορεύεται το να υπάρχει ε, μετεπιβίβαση ή μεταφόρτωση στα ανοιχτά πολλές φορές γίνεται μια τέτοια μεταφόρτωση πάρα πολύ μακριά από τους λιμένες. Πενταγουσίες κιλά που κάποιος ε, ψαρεύει στο, στον Πορντό και πάει μετά εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά να το πουλήσει. Αυτό γίνεται πάντως. Η, αυτή η μεταφόρτωση είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Γιατί αλλιώ θα έπρεπε κάποιο να κάθε τόσο να, να ξαναγυρίζει πίσω. Ε, Επομένω θα ήταν ε, οικονομικά σύμφορη μια τέτοια ρύθμιση. Υπάρχει μια αντίφαση γιατί λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι αρπαγορεύονται οι μεταφορτώσει στο άρθρο 13 και από την άλλη μεριά λέει, ή τουλάχιστον έτσι καταλάβαμε, έχουμε το 14 παράγραφο 3 εκεί που επιτρέπονται οι μεταφορτώσει. Αυτό λοιπόν που συνέταξε αυτέ τι διατάξει να μα τα εξηγήσει. Και λέει ότι ο πλοίαρχο ή ο εκπρόσωπό του επιτρέπεται να μεταφορτώσει κλπ. κλπ. Άρα λοιπόν, αλλού επιτρέπεται στο νομοθέτημα και αλλού απαγορεύεται η μεταφόρτωση. εκτο και έχει γίνει κάπου λάθο τη μετάφραση, δεν ξέρω. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο διαφωνούμε. Η ρύθμιση του άρθρου 14 παράγραφος 1 Εκεί που λέει θα πρέπει να υπάρχει μια προειδοποίηση τουλάχιστον 4 ώρων πριν μπει στο λιμάνι το πλοίο. Ε, αν όμως ε, ψαρέψει κάποιος μακριά από τα λιμάνια, δεν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι τέσσερις ώρες θα υπάρχουν για την ειδοποίηση. Αν όμως ε, γίνει στα χωρικά μας ιδιότητα σε κάποιο κόλπο της χώρας ας πούμε, ε, η αλίευση, γιατί θα κάτσει να περιμένει ο ψαράς τέσσερις ώρες για να κάνει την ειδοποίηση και να του επιτρέψουν να μπει στο λιμάνι. Εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτού του είδους η υποχρέωση να αφορά πολύ μικρότερο ε, χρονικό διάστημα. Μία, μία μισή ώρα θα αρκούσε αυτή η προθεσμία να ισχύει. Τέσσερι ώρες είναι υπερβολικό όταν κάποιος ψαρεύει ομένω στα χωρικά ύδατα της χώρα. Παρακάτω. Δεν συμφωνούμε για αυτό το περιθώριο του άρθρου 16. Μιλάμε για αυτό το 5% επίσης. Αυτό λέει ξεκίνησε σαν ρύθμιση αυτό το 20% από έναν κανονισμό του 83%. Ήταν 20% τότε όμως που ξεκίνησε αυτή η ιδέα του περιθώριου ανοχής και τώρα έπεσε στο 5% γιατί. Πολλές φορές εδώ έχουμε διαφορετικά αλλιεύματα, διαφορετικά είδη που είναι ανακατεμένα, επομένως αυτό το 5% ως περιθώριο μας φαίνεται πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ αυστηρό. Θα πρέπει να είναι επομένω πιο ψηλά το όριο ανοχής. Παρακάτω. Υπάρχει ένα θέμα εκεί σε αυτές τις διατάξεις για την εκμετάλλευση. Πρώτη της Κομισιόν που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. 0,30% είναι το ποσοστό εκμετάλλευσης. Ενώ προβλεπόταν 0,40% στο παρελθόν. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτό το 0,40. Αλλιώς υπάρχει εδώ κίνδυνος ε, ζημίας. Όσο αφορά το πρόγραμμα διαχείρισης υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Διακόπτη η πρόεδρος. Συγγνώμη σας διακόπτω. Παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί 12.30 θα πρέπει να κλείσουμε. Να τελειώσουμε τι συνεδρίε και θα πρέπει να μιλήσουν και άλλοι. Κάρα δύο πραγματάκια μόνο θέλω να σα πω ακόμα. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά το μέγεθο του αλλιεύματο δεν εμφανίζεται πουθενά, δεν ρυθμίζεται πουθενά σε αυτό το σχέδιο διαχείριση. Στο δε συμβουλευτικό ε, όργανο είχαμε πει ότι θα πρέπει για την ανοιχτή θάλασσα ε, για τις στράτες να είναι 50 κομμάτια ανά κιλό. Και προβλέπεται τώρα 90. Βλέπουμε επομένω ότι είμαστε πιο αυστηροί από όσα τώρα προβλέπονται. Ε, από αρχές Δεκεμβρίου μέχρι Φεβρουαρίου υπάρχει ε, η περίοδος απαγόρευσης αλίευσης, ε, αλίας. Τρεις μήνες είπαμε να, να γίνει αυτό, τόσο ώστε να μπορούν οι αλευτικοί πόροι να αναπαραχθούν. τέσσερα χρόνια. Είναι πέντε ελευθερικέ περίοδοι. Τόσο έχει κρατήσει αυτή η περιπέτεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα για τον ηλεκτρικό στόλο. Οπότε το 2010 επί τη βάση κάποιων ε, α, μελετών, επί τη βάση των προσδοκιών που ανοίγουν εξέλιξη της βιομάζης, επί τη βάση των οποίων οι επιστημονικοί οργανισμοί θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε την άνοιξη του 2010 επαναλαμβάνω, επί τη βάση των προσδοκιών για την αναπαραγωγή ε, της βιομάζης. Να συζητηθεί. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να είναι δυνατό αυτό που είπατε, λέει πρόεδρος. Παρακαλώ τώρα όλοι και άλλοι και άλλοι να μην μιλήσουμε μόνο πέντε λεπτά. Κύριε Ουριάρτε, έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Ήρθα εδώ για να σας μιλήσω για λίγο για το πώς εμείς από πλευράς άστε βλέπουμε αυτό το σχέδιο διαχείρισης. Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο, ήρθαμε σε επαφή με τους Γάλλους ε, ερευνητέ. Ε, οπότε δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να τα πούμε αναλυτικά μαζί τους, Θα είπαμε κάπως βιαστικά ό,τι προστάσαμε. Και θα ήθελα απλώ να σας αναφέρω ότι πρώτα πρώτα Είναι αξιόλογο αυτό το πρόγραμμα. Τα βασικά στοιχεία τα περιέχει, τα καλύπτει. Ξεκίνησε αυτή η διαδρομή το 2007, πέρασαν δύο χρόνια και ε, επομένω είχαμε πάρα πολύ μεγάλη πτώση και απομείωση των ε, αλληλευτικών πόρων. Χρειάζεται επομένω τώρα επιγόντω ένα τέτοιο πρόγραμμα, ούτω ώστε να σώσουμε του αλληλευτικού πόρου. Μέχρι τώρα δεν έχει σωστή διαχείριση και αυτό το τάκ των 3.000 που ήταν ε, φαίνεται αδόκιμο, ανεπαρκές και επίσης η διαδικασία ε, κατάρτισης του προγράμματος διακρίνεται από αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Ακούσαμε τα ΡΑΚ, ακούσαμε τους επιστήμονες, ακούσαμε την Κομισιόν. Οπότε και γι' αυτό σα λέω ότι θα πρέπει να δούμε ποιε ήταν οι διατάξει που διέπουν την εκμετάλλευση, αυτέ οι οποίε ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση αυτού του προγράμματο. Πώ δηλαδή διαμορφώθηκε το τελικό οριστικό κείμενο, η οριστική πρόταση αυτή, το οποίο παρουσιάστηκε εδώ, που βασιδευμένο σε κάποιε εκτεταμένε εξαντλητικέ μελέτε του Τεχνικού και Οικονομικού Συμβουλίου για την Ελία του οργάνου αυτού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επί τη βάση των στόχων που έχει τάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Ιούλιο με Ιούνιο είπαμε είναι η περίοδος της Αλίας που καλύπτει αυτά τα και κατόπιν κάποιων ε, αξιολογήσουν όσον αφορά του ελληνικού πόρου που έγιναν το Μάιο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε, να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο ε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Και έτσι να μπορέσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί για την χρήση των πληροφοριών, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη εκμετάλλευση των ελληνικών πόρων. Οπότε έτσι καταρτίστηκαν αυτοί οι κανόνε τη εκμετάλλευση. Έτσι έχω, φτάνουμε έτσι να δούμε πού είναι το maximum τη αλεία, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνο ε, για, το, για τους ελληνικούς πόρους, να μην κατεβαίνουμε κάτω από τα, τα όρια ανοχής της βιομάζας και είπαμε να μην πέσουμε κάτω από το 10%. Ε, αυτό είναι κάτι μια συντηρητικός υπολογισμός, μια που συζητήθηκε ε, πάρα πολύ όσον αφορά το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου για τη διαχείριση των πόρων. τώρα για τις νότιες περιοχές ε, ήταν πάρα πολύ προσεκτικό, είπε ότι εδώ πέρα ενέχονται, εδώ πέρα ενεδρεύουν πάρα πολύ σημαντικοί κίνδυνοι και επομένω είπαμε θα πρέπει να δούμε πώς θα φτάσουμε στην μεγίστη απόδοση χωρίς να διατρέχουμε κίνδυνο. Έχουν μέγιστες ποσοστώσεις και ελάχιστες ποσοστώσεις. Ε, αυτά ήταν επί τη βάση προτάσεων των Ελλήνων. Είχαμε τώρα κάποια στοιχεία τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη, όπως υπήρχαν κάποιε απαγορεύσεις τοπικές ή χρονικές σε σχέση με αυτά τα maximum και minimum ε, όρια επιτρεπόμενου ελλείμματο. Το CCTP δεν κάθισε να τα λάβει και αυτά υπόψη. Και αυτό δεν περιλήφθηκε σε αυτή την πρόταση για το διοικητικό πρόγραμμα. Έχουμε τώρα κάποια άλλα προβλήματα αυτή της πρότασης. Αυτή η προσέγγιση, ούτω ώστε να υπάρχει μια περίοδος Ιούλιο με Ιούνιο, όπω πρώτο το CCTP. Αυτό μα οδήγησε στο ότι σήμερα έχουμε πρόβλημα συγχρονισμού με την περίοδο αλίας. Και άρα υπήρξε πρόβλημα εφαρμογή του προγράμματος. Και τι κάνουμε, έτσι χάνουμε ευκαιρίες αλίευσης. Θα πρέπει να γίνονται οι, οι αλλαγές ή η η τα μεταβιβάσεις της ποσόστοσης με κάποιο άλλο τρόπο και λαμβάνοντας καλύτερα υπόψη την περίοδο αλίας. Άρα πρέπει να γίνει σε κάποια σημεία αναθεώρηση αυτού του προγράμματο διαχείρισης, επιδέχεται αλλαγές και έτσι να, αλλάξει, να αλλάξουν τα σημεία αναφοράς και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες προβολές. και να αλλάξει αυτή η ρήτρα αναθεώρηση που τώρα είναι τρίχρονη. Σας ξαναείπαμε ότι έχουμε έρθει σε κάποια συνεννόηση επιφανειακή με τους Γάλλου επιστήμονε και συμφωνήσαμε ω Επιστημονική Επιτροπή ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους λόγους που οδήγησαν στην πτώση των ελληνικών πόρων και άρα αυτό το πρόγραμμα διαχείρισης βασίζεται στο ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένα επίπεδα προσλήψεων. Και εισόδων στον κλάδο. Επομένως, έχουμε το άρθρο 5, παραγραφός 2, σε σχέση με τον υπολογισμό του μεγίστου αλλιεύματος. Εδώ η Επιστημονική Επιτροπή δεν μπόρεσε να διατυπώσει για την σημερινή βιομάζα μια πρόταση. δεν μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη κάτι τέτοιο στις προτάσεις που έγιναν. Το CCTV για τη Σαρδέλα είπε ότι θα πρέπει να έχουμε τα ωραία όσο γίνεται πιο χαμηλά και να γίνει αναθεώρηση στο 1 τέταρτον του περσινού τάκ. 7.000 τόνοι να είναι το ελάχιστο τάκ. ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη και ίσως να επαναδιατυπωθεί είναι να δούμε ξεκάθαρα υπό ποιες συνθήκες μπορούμε να έχουμε την αναθεώρηση του σημερινού προγράμματος. Πρώτον, αλλαγές στην επιστημονική γνώση. Κάτι το οποίο θα το πιστοποιήσει το ίδιο το CCTP. Άρθρο 6 ή άρθρο 22, εκεί θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για μια τέτοια αναθεώρηση. Ό,τι δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 6. Ακριβώς δηλαδή το CCTP το ίδιο να προτείνει ότι θα πρέπει να αλλάξουν ε, κάποια όρια ας πούμε, για τη βιομάζα. Να διατυπωθεί ας πούμε ότι δεν είναι βιώσιμο το επίπεδο της βιομάζας. και έτσι να φτάσουμε σε καλύτερη διαχείριση των ιδιωτικών πόρων μέσω αλλαγή των διατάξεων που αφορούν τις, ε, ε την εκμετάλλευση. Σας ευχαριστούμε για όσα μα είπατε, Πρόεδρε. Θα πρέπει να κλείσουμε σε πέντε λεπτά, γιατί έχουμε και άλλα θέματα σήμερα στη διάταξη. Η Guide. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των φορέων που ήρθαν να μας μιλήσουν. Πραγματικά άγγιξε την ουσία του προβλήματος. Και στέκομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Πάς στο τέλος, ότι έχουμε τέσσερα χρόνια, πέντε περίοδους αλίας που έχουμε κολλήσει χάνεται χρήμα, χάνονται απασχολήσεις, πάρα πολύ ε, ε, εξαρτώνται από αυτό το, κλάδο. Και μιλώ και για αυτούς που εξαρτώνται έμεσα, όπως ας πούμε αυτοί που κάνουν τα ψάρια κονσέρβες, όχι μόνο αυτοί που ψαρεύουν. Φυσικά και η απόρρευση ελίας είναι κάτι που το ζήτησαν πρώτοι οι ίδιοι ψαράδες. Με την φύλαξη του, τι θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ νομίζω όπως είπε και η κυρία Μπιλμπάου, θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει μια ρύθμιση σύντονη με αυτό το οποίο επιθυμεί ο κλάδος. Ξέρει η κυρία Μπιλμπάου τα θέματα. Να ληφθούν υπόψη τα αιτήματα του κλάδου επομένως και για τις προσαρμογές και για τον έλεγχο Έχουμε αυτέ όλε τι επιθυμητέ αλλαγέ που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό το κείμενο σαν προτάσει τη επιτροπή μα. Ωραία, όπω είπατε θα είμαι σύντομο και περιμένω πώς και πώς να ακούσω την Κομισιόν. Θα την υποστηρίξουν, Μακάρι. Τελικά να προκύψει από εδώ μία έκθεση που να υποστηρίζεται από όλε τι πολιτικέ πτέρυγε και έτσι να ωφελεί τον κλάδο των αλλιέων της Σαρδέλας και επιτέλους να λύσουμε το πρόβλημα που τους ταλανίζουν. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους ε, ομιλήσαντες για τα σχόλιά τους τα σχετικά με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Βιλμπάου, ετοιμάζουμε το κεφάλαιο αυτό για τον έλεγχο. Κάθε πληροφορία λοιπόν θα σας διατεθεί. με τις προτάσεις μας για τα διάφορα άρθρα. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω στον τομέα. Είχαμε διάφορες συνεδριάσεις την ομάδα μας και αντιλαμβάνομαι φυσικά την ε, σημασία που αποδίδεται στον έλεγχο. Θα πρέπει πιστεύουμε και στο μέλλον ε, να ε, έχουμε κανονισμό με συντονισμό και για τον τομέα της Αλίας στη Γαλλία αλλά και με την ε, Ισπανία, με τον Ισπανικό τομέα. Εκεί είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η έλλειψη ελέγχου πιστεύουμε είναι λόγος που μπορεί να οδηγήσει σε πολλές δυσκολίες και εδώ ακριβώς επισημαίνουμε τα προβλήματά μας. Ίσως λοιπόν οι 500 ετών να μην έχουν τόσο μεγάλη σημασία σε αυτή την περίπτωση. Γιατί λοιπόν να σταματήσουμε, γιατί σταματήσαμε να διαβιβάζουμε τα στοιχεία αυτά στην ε, επιστημονική ε, επιτροπή. Πρέπει να ρυθμίσουμε το πρόβλημα αυτό. των ζωντανών δολωμάτων. Ε, και στο κεφάλαιο του σχετικό με τον έλεγχο. Θα ήθελα να ακούσω τι έχει να πει πρώτα το Συμβούλιο. Και να δούμε από εκεί τι θα βγει. Υπολογίστε σε 40% περίπου βάσει τον κορώνα εκμεταλλεύση σε βιομάζα. Η Επιτροπή λοιπόν υπολογίζει τους ε, κινδύνους ε, σε πιο σημαντικούς από ό,τι περιμέναμε. Γι' αυτό προτιμάμε να είμαστε πιο ε, συνετοί και να περιορίσουμε τι προβλέψεις μας στο 30%. Για το μέγεθος του αλλιεύματος έχουμε να κάνουμε μάλλον με κεφάλαια σχετικά με τη ρύθμιση των αγορών. στο τέλος του έτους. Και νομίζω θα επανέρχομαι στο θέμα ως το θέμα του μεγέθους. Και θα ήθελα να πω ότι αφού δεν έχει γίνει πραγματικός διάλογος, συζήτηση για την διακοπή αυτή από το Δεκέμβριο στο Φεβρουάριο ε, μεταξύ των ηθικών. Δεν την αναφέραμε εμείς. Πιστεύουμε πάντως ότι το πρόβλημα και την επιστροφή στην έλλειψη συμφωνίας μεταξύ Ισπανών και Γάλλων και όταν βρέθηκε συμφωνία, ο τομέας μόνος του έλυσε το πρόβλημα. Όσο λοιπόν οι ειδικοί δεν μας έχουν δώσει πιστικά ε, επιχειρήματα ως προς τη χρησιμότητα αυτής της διακοπής είτε ως προς την ε, περίοδο της διακοπής είτε ως προς την ε, διάρκεια της τότε εμείς για αυτό το διάστημα επιφυλασσόμεθα. Άλλο στοιχείο, αυτόματη αναθεώρηση η οποία έχει σωματωθεί στο άρθρο υπαριθμών 6 από την στιγμή κατά την οποία η Συμβουλευτική Επιτροπή θα διαπιστώσει αλλαγή στον τρόπο χειρισμού του το αποθέματος ή αν αλλάξουν κάποια στιγμή τα δεδομένα θα πρέπει ενδεχομένως και να ξαναδούμε το σχέδιο, να το δούμε με διαφορετικό μάτι. Αυτά είχα να σας πω. Le agradezco, es que, es que de verdad a las doce y media los intérpretes se van y entonces... Στις 12.30 θα φύγουν οι δερμήνες. Επομένως, ε, όσο και αυτό να μην είναι τόσο βολικό, θα πρέπει να σας σταματάω. Ε, διότι θα πρέπει να τηρήσω τα ωράρια, τα ωράρια εργασίας των διερμηνέων. Ε, αλλιώς θα μπορούσαμε να κάτσουμε και να τα κουβεντιάσουμε. Κύριε Μπιλμπά, ένα λεπτάκι αν είναι δυνατόν. Muy rápido, pero... Αν μπορείτε να το μας τα πείτε γρήγορα. Εγώ. Δουλεύω, είμαι κοντά στον κλάδο και οπότε θα ήθελα από εδώ μέσα να βγει ένα κείμενο το οποίο να βρίσκει σύμφωνα όλα τα, τα κόμματα. Σας λέω για άλλη μια φορά, παρά το ότι αυτό δεν έχει κανένα πλαίσιο επίσημο, παρακαλώ η Κομισιόν να μας δίνει όσο και να δεν προβλέπεται πληροφορίες. Γιατί έχουμε αυτόν τον ε, κανονισμό που θέλει μέσα από το να περάσει το Συμβούλιο να προσέξουμε να μην βρεθούμε μέσα σε ένα παραλογισμό. Και θα καταλήξουμε τον Ιούλιο την τελευταία μέρα ε, πριν πάμε διακοπές, πριν, πριν κλείσει η ΟΚ, να, να δουλεύουμε στο γόνατο τελευταία στιγμή για ένα έγγραφο το οποίο είπαμε ότι καίει τον κλάδο. Έχουμε τέσσερα ε, άρθρα που αφορούν τον έλεγχο και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Παρακαλώ, δώστε μας ό,τι πληροφορίες χρειάζονται, τόσο ώστε αυτό που το κείμενο θα φτιάξω εγώ να, να έχει συνοχή, να έχει λογική, επί τη βάση και των ετοιμάτων του κλάδου, με κάποια διαδικασία, να προσέξουμε να αποφύγουμε το να βρεθούμε σε κατάσταση αντίφασης και παραλογισμού. Συνεργαστείτε μαζί μας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε τελικά να συμφωνήσουμε εδώ οι τα, θεσμικά όργανα για, την, για το όφελος του της Αλίας, για το όφελος της ΕΟΚ ε, και έτσι να, να έχουμε μια αξιοπιστία που πρέπει να έχουμε πρόεδρος. Α, στο σε τι, σε τι αναφέρεστε. Α, τώρα κατάλαβα, για τον ε, κανονισμό, τον ελεκτικό, εκεί αναφέρεστε. Α, μάλιστα, εντάξει. Και τώρα, προχωρούμε στο υπαριθμό 15 που είναι τα διάφορα. Θα ήθελε κάποιος κάτι να πει για τα διάφορα. Όχι, όχι κύριε κάτι άλλο θέλετε, εντάξει. Το τελευταίο τώρα. Πρόκειται για την ανακοίνωση σε σχέση με τι αποφάσει των συντονιστών. Σα έχω διανύμει το, σχετικό κείμενο. Αν δεν έχετε κάποια ένσταση, θα θεωρηθεί ότι οι αποφάσει εγκρίνονται. Για πάνω τόσο τελευταίο με τι μέρε διατάξει που είναι η μηνομία τη επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει στι Νοεμβρίου ή στι 3 μετά μεσημβρίων και στι 4 9 το πρωί. Πέρα συνεδρίασης.